Well, now that Mrs. Ruler is here, we can definitely start, because she is our most regular and persistent uh, attender of meetings. So... Κυρία Ρούλε, βλέπω είστε αφοσιωμένη στην, στις εργασίες μας. Ε, χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που είστε εδώ. Και η, η συγγήτριά μας είναι εδώ. Θα θέλω να καλωσορίσω και μια πάρα πολύ καλή ομάδα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Σαμπίντα Πρενιέζ είναι εδώ. Όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες σας είναι επίση παρόντες. Καλώς ήρθατε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ε, για την σημαντική μας γνωμοδότηση για τα ιατροτεχνικά προϊόντα. Μπορεί να τα ακούσατε, αλλά θα κάνω κι εγώ μια ανακοίνωση σημαντικά νέα και για όσους μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο γιατί κάποιοι το κάνουν. Και φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται πολύ ε, όσοι ανήκουν στην ιατροτεχνική κοινότητα. Η κυρία Νέβεν Νίμιτσα είναι επίτροπος ε, υποψήφιος ε, για την προστασία των καταναλωτών. Ε, νέο χαρτοφυλάκι από την 21η Ιουλίου. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ε, διορισμός, θα γίνει βέβαια και ακρόαση. Όσοι ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Νίμιατσα συγγνώμη, θα γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσωπικότητα. Προσπαθούμε όσο το συντομότερο γίνεται να οργανώσουμε την ακρόαση. Θα σας ενημερώσουμε για τη σχετική ε, ημερομηνία. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης θα ε, ήθελε να παραστεί στην ακρόαση. Θα ακούσετε βέβαια και περισσότερα, αλλά ήθελα να σας πω εγώ τα πρώτα νέα. Να περάσουμε τώρα στα σχέδια γνωμοδοτήσεών μας ε, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Διατροφικής Ασφάλειας, ασφάλειας των τροφίμων, η κυρία Νόρα Μπέρα, ε, είναι η δική μας εισηγήτρια, Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ για, ε, για την πρώτη έκθεση που αποτελεί αναδιατύπωση της τρέχουσας οδηγίας και επίσης για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro Χαίρομαι ιδιαίτερο που η κυρία Μπέρα εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Είναι εδώ για να μας παρουσιάσει τα ε, σχέδια γνωμοδότησής της και μετά ο καθηγητής Κορέα Ντεκάμπος που είναι σκιώδης εισηγητής για τους ε, ε, σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ να πάρει μετά το λόγο. κυρία Παρμανόβα δεν τη δεν τη βλέπω εδώ. Η κυρία Ρούλε μπορεί να την αντικαταστήσει ενδεχομένως. Ε, και ο κύριος Φόξ ε, δεν είναι εδώ, αλλά θα τον αντικαταστήσω εγώ. Να δώσω πρώτα το λόγο στην ε, κυρία Μπέρε να μας παρουσιάσει τις ονομοδοτήσεις της. Merci, Monsieur le Président, euh, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς ε, να καλωσορίσω την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και τη Γραμματεία. Επειδή ο χρόνος ε, που έχουμε στη διάθεσή μας παρά το περίπλοκο του ζητήματος, ε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και συνοπτική. Όσον αφορά τώρα τις εκθέσεις μας, την έκθεσή μου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μιλήσω για το πεδίο εφαρμογής. Μου φαίνεται σημαντικό να διευκρινίσω το θέμα τα, των αισθητικών ε, ε, ιατροτεχνικών προϊόντων που δεν έχουν δηλαδή φαρμακευτικό σκοπό αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα ε, έγχρωμη φακή οράσεως, ε, φακή επαφής. νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε έναν θετικό κατάλογο ε, δεν θα ήταν καλό να είχαμε συγγνώμη έναν, καλό, έναν θετικό κατάλογο ε, γιατί θα υπήρχε το πρόβλημα της ε, διεξοδικότητας, υπάρχει το θέμα για παράδειγμα της ε, ραδιοσυχνότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται αν είχαμε ένα τέτοιο κατάλογο ενώ θα έπρεπε. Έχουμε λοιπόν έναν ειδικό ορισμό που θα έπρεπε να καλύπτει όλα τα προϊόντα που έχουν τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου ιατροτεχνικού προϊόντος. Θα ήθελα να παρουσιάσω τον ορισμό αυτό για να εξασφαλίσω την συνοχή όπως επίσης κάποια προϊόντα όπως για παράδειγμα τα ε, σκουλαρίκια να τα ε, αποκλείσω πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες ταξινόμησης. Ε, γνωρίζετε ότι στο παράρτημα 7 υπάρχουν οι κανόνες 19 και 21, πρέπει να τους προσαρμόσω για να δείξω ότι κάποια προϊόντα για την ώρα δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο και δεν θα έπρεπε να ε, διέπονται από πολύ βαριέ διαδικασίες. Και αναφέρομαι σε κάποια ε, πρόσθετα, οδοντικά ή σπρέι γιατί ρινικά σπρέι, ε, τα οποία δεν υπήρχε λόγος να περάσουν τέτοιε διαδικασίες. Ε, όμως πιστεύω ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση επαρκής και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να διαγραφεί ο κανόνας αυτός. Πρέπει να είμαστε σαφείς ή πρέπει να πούμε ότι ανταποκρίνεται κάτι σε ένα προϊόν, στον ορισμό ενός προϊόντος ιατροτεχνικού προϊόντος, δηλαδή και να, υπάρχει, να μην υπάρχει κίνδυνος, ε, δηλαδή καλύπτεται από την κατηγορία 3 όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό. Ή υπάρχει ορισμός του φαρμάκου και σε αυτή την περίπτωση ε, διέπεται από την οδηγία για τα φάρμακα. Αν δεν υπάρχει όμως ε, ιατρικός στόχος, κανένα από τα προϊόντα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται ιατροτεχνικά ε, προϊόντα και πρέπει να διέπονται από την σχετική νομοθεσία. Ε, όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα τα ιατροτεχνικά προϊόντα και τι θα πρέπει να καλύπτει, το επίπεδο του κινδύνου είναι που μας ενδιαφέρει. Να δούμε τώρα πώς θα το οριοθετήσουμε αυτό. Να μην υπάρχουν ε, διαφορές στην ερμηνεία όσον αφορά το, το καθεστώς των προϊόντων αυτών μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα ε, στο άρθρο 15 της πρότασης. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια πραγματική γκρίζα ζώνη σε σχέση με την επεξεργασία. Ε, ένα προϊόν μπορεί να, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να, πολλές φορές να έχει ένα κύκλο ζωής ή μπορεί να έχει μία και μοναδική χρήση, οπότε ε, δεν μπορεί να, να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Υπάρχουν όμως όλο και περισσότερα προϊόντα ε, που η ετικέτα τους λέει ότι είναι μοναδικής χρήσης, μίας και μόνης χρήσης, όμως θα μπορούσαν να ε, ξαναχρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, σε ορισμένα νοσοκομεία γίνεται τέτοιου είδους εκ νέου χρήση. Ε, και μιλάω για παράδειγμα για τα ηλεκτρο... τα ηλεκτρόδια, τους καθετήρες. Ε, Μπορούμε βέβαια να χτενίσουμε λίγο τον ορισμό αυτό, να πούμε τι ακριβώς είναι επιστημονικός ορισμός. Μπορούμε να περιορίσουμε ε, κάτι τέτοιο μόνο στα προϊόντα ε, για τα οποία χρειάζεται μια τέτοιου είδους διευκρίνηση. Δεν είναι πάντοτε ε, απαραίτητο αυτό. Για παράδειγμα ένα προφυλακτικό δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνει αυτή η οριοθέτηση ε, προϊόν μπορεί να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, να είναι μία και μοναδική χρήση εκτός εάν ε, καταδεικνύεται κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί λοιπόν τότε ο, ο κατασκευαστής να γράφει ότι ε, είναι μίας χρήσεως, αλλά προορίζεται για μία και μόνη χρήση, δηλαδή συστήνει μία ε, μοναδική χρήση, όπως για παράδειγμα για το καφετήρα, χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα εκ νέου χρήσης, ενώ υπάρχει περίπτωση πολλαπλής χρήσεως, ε, όπου αναφέρεται πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για πόση διάρκεια ε, κλπ. Όσον αφορά τώρα αυτόν που το ξαναχρησιμοποιεί, μια εταιρεία, ένα νοσοκομείο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η νέα χρήση γίνεται με ασφαλή τρόπο και βεβαίως να υπάρχει μια νομική ευθύνη για το προϊόν. Ε, πρέπει λοιπόν οι ευθύνες να είναι ε, σαφέ, σαφείς και να μην υπάρχουν υπερβολικές υποχρεώσεις που να βαρύνουν τον κατασκευαστή. Όσον αφορά τώρα την τοποθέτηση στην αγορά επικίνδυνων προϊόντων και μιλάω για το άρθρο 44. Πρόκειται για ένα από τα πιο επίμαχα σημεία της πρότασης αυτής. Νομίζω συμφωνούμε ότι το σύστημα έχει κενά ε, και ότι βεβαίως επιδέχεται βελτιώσεων επειδή υπάρχει μαζική εισαγωγή θεραπευτικών όλο και περισσότερο καινοτόμων θεραπευτικών ε, προϊόντων ε, όπως για παράδειγμα όλα τα προϊόντα που, πιτρέ, χρειάζεται, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνει χείριση ανοιχτή καρδιάς η σταθεροποίηση της πονδυλικής στήλης κάτι το οποίο σημαίνει ότι μερικέ φορές δεν έχουμε αρκετή επιρρογνωμοσύνη για να δούμε, ε, να αξιολογήσουμε τις κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει από τον κατασκευαστή. Ε, όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο έλεγχος αυτός θα γίνει με εναρμονισμένο τρόπο σε 80 ε, κοινοποιημένους διαφορετικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Χρειάζεται μία μόνιμη αποτελεσματική λύση μεταξύ της κεντρικής αδειοθότησης τοποθέτησης στην αγορά και του συστήματος του τρέχοντος που βασίζεται αποκλειστικά τώρα στην πιστοποίηση από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Άρα προτείνω ένα εναλλακτικό σύστημα. Εκτός από την ενίσχυση των απαιτήσεων που ισχύουν για τους κοινοποιημένους οργανισμούς προτείνει η Επιτροπή. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές, τέλος πάντων συστάσεις καλής πρακτικής για την κλινική αξιολόγηση, για να αντιμετωπίσουμε ε, τις διαφορετικές αξιολογήσεις των κοινοποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή αυτές, ε, υπάρχουν αυτές οι ευρωπαϊκές συστάσεις, θα έχουμε την εγγύηση ότι γίνεται ε, έλεγχος ομοιόμορφος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, θα υπάρχουν πάνελ εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αξιολογήσουν τα πιο ευαίσθητα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές. Πρότεινα να επικεντρώσουμε στις κατηγορία, στην κατηγορία 3 τις εμφυτεύσιμες ιατροτεχνικές συσκευές, ε, ε, ε, το προϊόν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό ε, αποδεκτό υπό προϋποθέσεις, ε, τροποποίησης ε, της συνταγής, του τρόπου εμπορευματοποίησής του ή θα μπορούσε να απορριφθεί. Πέρα από αυτό, ε, οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα έχουν ως καθήκον να ε, ορίσουν αυτούς τους οδηγούς καλής κλινικής πρακτικής που μας λείπουν για αυτά τα ιατροτεχνικά προϊόντα τα πιο επικίνδυνα. Ε, αυτή τη στιγμή βέβαια έχουν αξιολογηθεί τα προϊόντα αυτά και βεβαίως υπάρχουν σχετικά στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα αυτά μετά δεν θα χρειάζεται να περνά συνεχώς έλεγχο το προϊόν και θα μπορούσε να ακολουθεί την κλασική διαδικασία μέσω ενός κοινοποιημένου οργανισμού. Το σύστημα θα σήμαινε ε, ότι κάποια προϊόντα θα περνούσαν, θα θεωρούνταν εγκεκριμένα, όμως θα, θα, θα βασιζόταν στη συνέχεια σε πιο καινοτόμα για να πλαισιωθούν κάπως τα συστήματα τα ευρωπαϊκά, να βελτιωθεί ο έλεγχος των, των κοινοποιημένων οργανισμών ε, για τα επικίνδυνα προϊόντα, χωρίς να είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ ε, παγιωμένο αυτό το σύστημα ε, και θα παρέμενε στο πνεύμα της νέας προσέγγισης. Και υπό το πνεύμα αυτό εγώ σας πρότεινα τη δυνατότητα ενός επιστημονικού συμβουλίου εκ των προτέρων ε, για όλους όσους ε, για όλους κατασκευαστές που αφορά αυτό το θέμα για να δούμε καταρχάς τι περιμένουμε από την κλινική αξιολόγηση του προϊόντου του ειδικότερα όσον αφορά ε, το κομμάτι πριν αλλά και μετά από την εμπορευματοποίηση. Πρέπει λοιπόν να επαχρυπνούμε, να μην εισάγουμε οργανισμούς που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα ενός πολύ καινοτόμου ανταγωνιστικού ε, τομέα ε, με χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας για την Ευρώπη και πιστεύω, πιστε, πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι για ένα, χρο, ένα αριθμό επικίνδυνων ιατροτευτικών προϊόντων η αξιολόγηση από κοινοποιημένου οργανισμούς δεν είναι παρκής και γι' αυτό η προσέγγιση μου έχει ε, νομίζω πιθανότητες να θεωρηθεί καλός ε, συμβιβασμός. Για τους ε, in vitro, για τα in vitro ιατροτεχνικά προϊόντα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και γι' αυτό προτείνω μια υποχρέωση εγγύηση των κατασκευαστών για να καλύψουν ενδεχόμενο κίνδυνο ανεπάρκειας βλάβης των προϊόντων τους. Νομίζω ότι πρέπει να ε, πούμε ε, τι θα μπορούσε, τι θα μπορούσε να καλύπτει μια τέτοιου είδους ασφάλεια. Πιστεύω επίσης ε, ότι οι ευθύνε πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να μην υπάρχει κατακαιρματισμός τους, κάτι το οποίο ουσιαστικά θα έπλητε τη συγκεκριμένη πρόταση. Κάτι ακόμη τώρα για τα διαγνωστικά προϊόντα in vitro, βεβαίως υπάρχουν κάποια παράλληλα στοιχεία με, το, με την προηγούμενη μου γνωμο, με την άλλη μου γνωμοδότηση που μόλις σας παρουσίασα. Νομίζω ότι πρέπει να πλαισιώσουμε καλύτερα ε, ε να, ξέρουμε δηλαδή την, ε, τα, τα τεστ ε, DNA αν θα έπρεπε να τα συμπεριλάβουμε αν δεν έχουν ιατρικό στόχο αλλά ε, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή ρύθμιση. Θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό ακριβώς το σημείο πριν εγώ ε, προτείνω διατάξεις, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε ε, αρκετή έρευνα σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα δουλέψατε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα γιατί έχετε καταθέσει και ένα σωρό τροπολογίε. και σας ευχαριστώ που μας δείξατε πόσο ειδικοί είστε για το θέμα. Έχουμε χρόνο για συζήτηση ε, και είναι καλό που μας το εκθέσατε έτσι αναλυτικά. Έχουμε εδώ τους Κιώδης, τον Αντώνιο Κορέιο Κάμπος, ε, την Αντώνη Παρμανόβα και την ε, Χάιδη Ρούλε. Ο Αντώνιο Κορέιο Κάμπος. Ευχαριστώ Μάλκομ. Πρέπει να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Νόρα Μπέρα, όπως το είπατε κι εσείς, διότι μπόρεσε να μεταφέρει την προηγούμενη επαγγελματική της γνώση, την πείρα της, για να προετοιμάσει μια πολύ σημαντική και ουσιαστική ανάλυση για αυτή την έκθεση. Τώρα θα τα πω αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία για την Έγκριση Τεχνολογικών ε, Προϊόντων έχει καλά χαρακτηριστικά ευελιξίες και ταχύτητας που θα πρέπει να διατηρηθούν. Το σύστημα ευνοεί την ιατρική καινοτομία και την γρήγορη πρόσβαση των ασθενών ε, στις θεραπείες, στις αγωγές αυτές. Ε, θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίσουμε τη ευάλωτα σημεία όπως η κλινική αξιολόγηση των καινοτόμων για το τεχνολογικών προϊόντων ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των ασθενών. Ωστόσο, ένα σωρό προϊόντα ε, έρχονται στην αγορά από ό,τι καινοτόμα φάρμακα. Και εξάλλου για τα τεχνολογικά προϊόντα και τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι πολύ διαφορετικά στη δράση τους ε, στο σώμα, στο ανθρώπινο σώμα και αυτές οι διαφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας τους. Αυτή η ε, διαδικασία δεν πρέπει να επιβαρυνθεί για να μην επιβαρυνθούν οι μικρές καινοτόμε εταιρείε, χωρίς να προσφέρουμε και περισσότερη ασφάλεια στους ασθενείς από ότι ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν να δοθεί στη εποπτικός ρόλος στο ε, συντονιστικό όργανο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θεωρούμε ότι οι προτάσεις της εισηγήτριας ε, κάπως είναι υπερβολικές ε, όσον αφορά την κεντρική διαχείριση που προτείνεται. Βεβαίως ε, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συμβιβαστούμε. Προτείνουμε ωστόσο να γίνουν κάποιες αλλαγές στο ενεργασία των και κοινοποιημένων οργανισμών, ώστε αυτή να είναι πιο απαιτητική. Όσον αφορά τους κοινοποιημένους οργανισμούς, εμείς ε, υποστηρίζουμε την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους εθνικούς ε, ρυθμιστές, ώστε να μπορούν να ελέγχουν λεπτομερώς τις δραστηριότητες των κοινοποιημένων οργανισμών. Χρειάζεται επίσης περισσότερη διαφάνεια για την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης των ιατροτεχνολογικών ε, ε, προϊόντων. Θα πρέπει να ενημερώνονται τα κοινοποιημένοι οργανισμοί, αλλά δεν θα πρέπει αυτοί να εγκρίνουν οποιοδήποτε κλάση προϊόντος. Θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια για τους κοινοποιημένους οργανισμούς, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη προσπάθεια εποπτείας και ελέγχου. Για τις κλινικές μελέτες, ε, παρά το γεγονός ότι οι κλινικές μελέτες για τους ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι, διαφορετικές από ό,τι κλινικές ε, δοκιμές για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Μπορούμε ωστόσο να ενισχύσουμε τις προδιαγραφές για τις κλινικές ε, μελέτες. Και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό, αλλά γνωρίζουμε πως υπάρχουν ε, δυσκολίες στο να γίνονται ε, μελέτες πριν την εμπορία ενός προϊόντος για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά του. Αυτό ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο να γίνει. Τώρα, η ε, πανεπεξεργασία ή ε, ε, προϊόντων μιας χρήσης. Αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο, όπως ήδη τονίστηκε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η πανεπεξεργασία προϊόντων μιας χρήση θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα και ότι η προστιθέμενη αυτή χρήση θα επιτρέπεται από τον αρχικό κατασκευαστή και θα εξετάσουμε και πάλι την πρόταση αυτή πριν προτείνουμε αλλαγές. Για την εποπτεία και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ε, είναι ένα από τα βασικά ζητήματα αυτής της έκθεσης. Στηρίζουμε ε, έγκυρη και πιο εντατική παρακολούθηση ώστε να έχουμε θετική ε, εικόνα και διαφάνεια και ανιχνευσιμότητα. Ε, ε, ξαφνικές επισκέψεις, εφόδους στους κατασκευαστές ε, με βάση ένα προκαθαρισμένο κατάλογο προδιαγραφών. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρόσβαση σε στοιχεία πριν προεμπορίας και μετά εμπορίας των προϊόντων. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και για τα στοιχεία που δίνει ο χορηγός πριν από την έγκριση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο απόρριτα εμπορικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων ε, ε, μέσων και είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο αλλά και για τους ερευνητές. Είναι ένα μέσο για την καλύτερη γνώση των επιδόσεων των προϊόντων των ιατροτεχνολογικών. Ε, αυτή είναι, Πρόεδρε, μια πολύ σημαντική και δύσκολη υπόθεση, μελέτη και εγώ ο κανονισμός είναι πολύ δύσκολος. Χρειάζεται να δουλεύει δουλέψουμε πολύ ακόμα πάνω σε αυτόν. Εδώ είμαστε ακόμα... Έχουμε απλά μια γνωμοδότηση να συντάξουμε, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε η τελική απόφαση να είναι ή κατάλληλοι στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, είναι καλό να έχουμε τόσο πολλούς ε, καλούς εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή μας και ξέρω πως και η κυρία Παρβάνοβα γνωρίζει εις βάθος το θέμα και της δίνω το λόγο. Έχουμε ένα σωρό χρόνο έτσι κι αλλιώς, γιατί το επόμενο μας ε, σημείο προβλέπεται για τις 4. Για μια φορά μπορώ να σας πω, μπορείτε να μιλήσετε με την ησυχία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, το θέμα είναι τόσο περίπλοκο και τόσο σημαντικό και πραγματικά λυπούμε που δεν είχαμε ε, την τύχη να έχουμε τόσο καλούς ε, και εμπειρογνώμονες συζητητές σε άλλα θέματα, όχι μόνο σε ανταγωνισμό με την Εύη να μπορούμε να δουλέψουμε, αλλά σε συνεργασία μαζί της. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω μάλλον την εισηγήτρια που διευκρινίζει τις αρμοδιότητες της Ένωσης ε, ώστε να αποφευχθούν ε, συγκρούσεις με τη επιτροπή μα τη Αρμοδιότητα, με συγχωρείτε, ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε διαμάχη με την Επιτροπή περιβάλλοντο. Ε, το θέμα αυτό προκαλεί σκληρέ έντονε συζητήσει στο σώμα, ανάμεσα στι επιτροπέ, αλλά και ανάμεσα στι πολιτικέ ομάδε και του διάφορου πυρογνώμονε ευρωβουλευτέ και σε εθνικό επίπεδο. Και ιδιαίτερα όσον αφορά το κατά πόσο θα πρέπει να ενισχυθούν ή όχι και με ποιο τρόπο η διαδικασία προηγούμενης αξιολόγησης πριν δηλαδή τη διάθεση στην αγορά. Η συγγήτρια της ΕΝΒΗ προτείνει κεντρική έγκριση ή μάλλον διαδικασία κεντρικής έγκρισης για την κλάση 3 ε, τέτοιων προϊόντων πριν τη διάθεση στην αγορά. Η δική μας πρόταση είναι παρόμοια και όποια και αν είναι η τελική λύση, πιστεύω πως η πρόταση της κυρίας Μπερά ε, να κινείται πιο προς μια συμβιβαστική ε, λύση αν ε, μιλήσουμε για δεσμευτική γνωμοδότηση του συντονιστικού οργάνου ιατρικών συσκευών για ίσως θα πρέπει να δούμε λοιπόν μήπως έτσι μπορέσουμε να βρούμε μια ε, συμβιβαστική λύση. Εν γέννη χρειάζεται να υπάρξει έτσι ενισχυμένη προσέγγιση. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ιδιαίτερα στον κλάδο αυτό ότι μια πιο κεντροποιημένη και ενισχυμένη διαδικασία με κοινοποιημένες ε, αξιολογήσει μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Εγώ ωστόσο θα ήθελα να τονίσω ότι η ε, ασφάλεια των ασθενών είναι πολύ πιο σημαντική, ιδιαίτερα αν δει κανείς το μακρύ κατάλογο περιπτώσεων και προϊόντων που δεν είχαν εγκριθεί από την ε, ε, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΙΠΑ και αργότερα αποσύρθηκαν από την αγορά ενώ είχαν προκαλέσει πολλά προβλήματα ακόμα και θανάτους. Είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έχει ευθύνη, φέρει ευθύνη για τη δημόσια υγεία ενώ οι κοινοποιημένοι οργανισμοί στην Ευρώπη δεν φέρουν τέτοια ευθύνη. Και αυτό σημαίνει διαφορά όσον αφορά την ασφάλεια. Όσο, ε, με την κυρία Μπερά θα πρέπει μάλλον να το συζητήσουμε όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού, την σύσταση των κοινοποιημένων οργανισμών, ώστε αυτοί να ενισχυθούν. Γιατί μέχρι στιγμής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξωτερικοί σε πράγμα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και σύγκρουση συμφερόντων καθώς και ως προς τον εντοπισμό της σύγκρουσης συμφερόντων κάποιες φορές. Πιθανότατα θα πρέπει να ενισχύσουμε την διαφάνεια. Και στη συνέχεια όσον αφορά την σύσταση των στοιχείων ε, για την αξιολόγηση πριν τη διάθεση στην αγορά, θα πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητά της, να το συζητήσουμε και να το προσθέσουμε και όχι μόνο να μείνουμε στην ασφάλεια και στην απόδοση, αν και πιστεύω ότι η απόδοση θα πρέπει να καθοριστεί καλύτερα γιατί μέχρι στιγμή δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό. και μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην ερμηνεία. Ένα άλλο θέμα που πιστεύω ότι μπορούμε να προτείνουμε για να βελτιώσουμε την ασφάλεια είναι <laughs> η απόδειξη της προστιθέμενης αξίας. Όχι μόνο ανάμεσα στην προηγούμενη έκδοση της ίδια, του ίδιου προϊόντος, αλλά και σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα, πράγμα που θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αργότερα για την αποζημίωση των προϊόντων αυτών και για την εφαρμογή, την χρήση τους στα νοσοκομεία. Και πάλι τώρα για το σκοπό της ε, αξιολόγησης πριν τη διάθεση στην αγορά και ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις επικάλυψης ε, για τους κοινοποιημένου οργανισμούς ή οποιαδήποτε διαδικασία επιλέξουμε για την ενίσχυση του ρόλου των κοινοποιημένων οργανισμών θα ήταν ίσως χρήσιμο τα προϊόντα κλάσης 3 να μην εξετάζονται σύνολα αλλά να χρησιμοποιηθούν κριτήρια και να δημιουργηθεί μια υποομάδα κλάσης 3 που θα ήταν πιο κατάλληλη για μια τέτοια διαδικασία. ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για εμφυτεύματα εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε περισσότερο για λόγους ασφάλειας. Επίσης για την, ε, την έγκριση πρώτης διάθεσης στην αγορά, θα πρέπει εδώ να συμφωνήσουμε για όποιο σύστημα είναι, θα πρέπει αυτά να καταγράφονται στο Μητρό και μετά να αυξάνονται οι έτσι δυνατότητες για την ανιχνευσιμότητα, για να μην αναφέρουμε τον αριθμό περιπτώσεων, περιστατικών που δημιουργούν πρόβλημα λόγω της έλλειψης βάσεων δεδομένων και εργαλείων για την ανείχνευση των προϊόντων αυτών. Συμφωνώ επίσης με τον συνάδελφο ότι τα κριτήρια και οι ορισμοί για τις καινοτόμες ε, ε, για τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρειάζονται και θα πρέπει να προσθεθούν στην πρόταση. Ένα κρίσιμο θέμα για, για τα τεχνικά κριτήρια είναι ότι κατά τη γνώμη μου για τα ουσιαστικά κριτήρια για να μην υπάρχει ασάφεια και είναι καλύτερο να, είμαστε, να, να, περιλαμβάνονται στον κανονισμό, ενώ για τα δευτερεύοντα κριτήρια να μείνουμε στην κατεξιδότηση πράξη. Έπειτα, το επίμαχο θέμα της επανεπεξεργασία. Δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη αυτή η πρακτική στην Ευρώπη. Είναι αρκετά επίμαχο το θέμα και ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά είναι ένα ολόκληρο κλάδος ε, μπορεί να σκεφτούμε να νομοθετήσουμε εκεί χωριστά. Μέχρι στιγμής όμως πιστεύω πως υπάρχει επικάλυψη. Η ε, παραπλανητική ενημέρωση όσον αφορά τη μια χρήση ή την επανεπεξεργασία. Βέβαια, η μια χρήση και η επανεπεξεργασία δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την ευθύνη, τη λογοδοσία κτλ. κάτι αργότερα πάει στραβά. Αν όμως κάτι φέρει το σήμα μιας χρήσης, θα πρέπει να μένει μια χρήση. Η επαναπεξεργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο σε περιπτώσει όπου είναι αποδεδειγμένο πω είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όχι εκεί όπου αναφέρεται συγκεκριμένα πως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Έπειτα, πιθανότατα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της κατάχρησης της μιας χρήσης της ηθικής μάλλον ε, κατά, κατάχρησης των προϊόντων μιας χρήσης. Υπάρχουν όλα ένα και περισσότερες περιπτώσεις και πρέπει να αναλυθεί το γεγονός ότι για εμπορικούς σκοπούς κάποιες φορές ε, ο κλάδος χρησιμοποιεί διαφορετικές εμπορικές εμ, τεχνικές ώστε να... υπάρχουν διαφορετικοί ε, διακόπτε ή διάφορα εξαρτήματα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε το σύνολο να συνδέεται με έναν κατασκευαστή, αλλά και με τα φάρμακα που περνούν μέσα από το συγκεκριμένο προϊόν. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε όμως με επαναπεξεργασία. Ούτε με το κατά πόσο είναι μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων αν αυτό αποστηρωθεί δηλαδή. Καλύτερος τρόπος είναι να το χωρίσουμε σε ένα διαφορετικό νομοθέτημα αυτό το θέμα, γιατί αν δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και τις θέσεις των κρατών μελών, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι τα περισσότερα από αυτά θα συμφωνήσουν να ανοίξουν αυτό το θέμα μέσω του εδώ της νομοθεσίας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι εγώ, και ο Σκιάδη, εισηγήτρια και σίγουρα και οι άλλοι συνάδελφοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την εισηγήτρια και να διευκολύνουμε και την εργασία της Επιτροπής ΕΝΒΗ ώστε να υπάρξει καλή συνεργασία ανάμεσα στις Επιτροπές τις δύο και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μας οι μας, όλοι προβληματισμοί της ΙΜΚΟ θα ληφθούν ε, υπόψη. Δεν είναι πάντοτε δυνατό αυτό, αλλά θα μπορέσουμε νομίζω να υπερασπιστούμε τη θέση μου και έχουμε εξαιρετική εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed. Again, some... Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ πολύτιμα αυτά τα σχόλια, η κυρία Ρούλε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και η κυρία, ιδιαίτερα την κυρία Παρβάνοβα. Με βοήθησε πάρα πολύ εγώ ειδικό δεν είμαι σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν άλλοι τομείς που είμαι πιο εμπειρογνώμων από αυτό. Και είπα όμως από την περασμένη φορά ότι ορισμένα τμήματα αυτών των εκθέσεων υπερβαίνουν κατά πολύ τη δική μας αρμοδιότητα και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αρμοδιότητά μας και να περιοριστούμε σε αυτή. Έκανε τροπολογίες η κυρία Παρβάνοβα. Όχι η συγγήτρια, συγγνώμη, διορθώνει η κυρία Ρούλε, μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν αυτές οι αλλαγές καλύπτονται από τη μελέτη σκοπιμότητας, διότι δεν την έχω καταλάβει ακριβώς αυτή την ιστορία. Και θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Παρβάνοβα για την επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση. Αν δεν απατώμε πριν από τέσσερα χρόνια, ίσως και παραπάνω, κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση Ε, και είπαμε ότι υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη και δεν ξέρω αν υπάρχει καμία δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ε, θα προτιμούσα να το ξεχωρίσουμε γιατί μόνο προβλήματα θα έχουμε με το Συμβούλιο και εγώ επιθυμώ ο κανονισμός να εγκριθεί όσο γίνει το συνομότερο. Εάν τα τσουγκρίσουν πάλι στο Συμβούλιο για να το πω έτσι για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων ε, θα έχουμε πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω και το Συμβούλιο. Αν διευρύνει το πεδίο εφαρμογή, είμαστε εντάξει, καλύπτεται αυτό από τη μελέτη σκοπιμότητα ή χρειάζεται κάτι άλλο. Και τι γίνεται με τη δομή και τη διάρθρωση που προτείνει και η συγγήτρια τώρα, αλλά και η άλλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ, περιβάλλοντος, την ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει να πει τίποτα σχετικά να το σχολιάσει. Ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω τώρα τον εισηγητή, το σκιώδη εξ του κυρίου Φόξ και είναι και τεχνικά αυτά ε, που μας έχει δώσει. Μια άτυπη δική μου παρατηρησία, ε, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Υπάρχει μεγάλη πίεση ε, ε, στους προϋπολογισμούς της ε, υγείας και θέλουμε να δούμε και από τις δημόσιες προμήθειες ε, τι μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ποιες είναι οι παναχρησιμοποιούμενες λοιπόν τέτοιες συσκευές ή συσκευάσματα. Θα, θα τα πει και ο κύριος Φόξ αυτά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να το αφήσουμε απαραίτητα στον κατασκευαστή αυτό, δηλαδή να ορίζει αυτός που φτιάχνει ένα προϊόν αν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή ε, να πεταχτεί παρόλο που δεν υπάρχει προφανής και ε, πρόδειλος ιατρικός λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Φόξ καλωσορίζει την πρόταση αυτή και την νομοθεσία και πιστεύει ότι θα αυξήσει την ποιότητα όσο και την ασφάλεια των ιατρικών τρο τεχνολογικών σκευασμάτων και των in vitro ε, υλικών ε, και θα βοηθήσει ε, και στην καινοτομία και στην ενημερωμένη επιλογή των καταναλωτών. Ανησυχεί πολύ όμως με άλλα θέματα που αφορούν τις τροπολογίες και τα πόσο βοηθούν τον καταναλωτή, γιατί η δική μας ε, σκοπιά αυτή είναι η προστασία των καταναλωτών. Υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυρίας Μπερά για ε, τον ορισμό του ενεργού ε, σκευάσματος υλικού, δηλαδή όχι σύριγγες και τέτοια αναλώσιμα, αυτά ξερούνται και γάζες. Υπάρχει μια ομάδα συντονισμού ε, συμφωνεί με τη διαφάνεια και τη μεγαλύτερη πληροφόρηση για τις συσκευές αυτές και τα ε, προϊόντα για να ξέρουν και οι κατασκευαστές που να κινούνται. Ωστόσο, διαφωνεί με την ε, γνωμοδότηση σε διάφορους τομείς ο κύριος Φόξ και θα σας τα πει σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ίδιος στη συνεδρίαση των σχεδόν Υποστηρίζει ορισμένα προϊόντα που εμφυτεύονται ε, στο σώμα, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί ένας γενικός ορισμός για όλα τα προϊόντα. Συμφωνεί με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράρτημα που θα απαριθμεί τα προϊόντα αυτά. Επίσης υποστηρίζει ε, την αρχή ότι ένα σκευασμό θα είναι είτε μιας χρήσεως είτε επαναχρησιμοποιούμενο. Δεν θα είναι τα δύο. Ε, και μπορεί ε, να μην επαναχρησιμοποιείται για λόγους προφύλαξης αναπριών όταν δεν υπάρχει ε, ιατρικός λόγος ή απόδειξη. Το άρθρο 43 θα προκαλέσει επιπλέον κόστος επικαλύψεις και διπλοδουλειές χωρίς να δίνει επιπλέον ασφαλιστικές δικλίδες για τους καταναλωτές. Και οι προτινόμενες αλλαγές εντείνουν τα προβλήματα αντί να τα επιλύουν. Κατά την άποψή του θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των σωμάτων που δέχονται τις αναφορές και τις κοινοποίησεις για να μπορούν να αντιδρούν και να έχουν γρήγορα πρόσβαση οι καταναλωτές σε καινοτόμες συσκευές και σκευάσματα που δικαιούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα τα in vitro ιατροτεχνολογικά ε, προϊόντα θα πρέπει και πάλι να ε, διευκρινιστούν κάποια θέματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογή ε, και τις δοκιμές και τα πειράματα που γίνονται ε, στα νοσοκομεία. και για τα συσκευές in vitro της κατηγορίας α έως δέλτα και για σπάνια νοσήματα. Και αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις ε, σε ζωτικές υπηρεσίες διάγνωσης. Ε, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μελέτη αντικτύπου είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε για τα επιστημονικά ούτε για τα ε, οικονομικά ζητήματα. Και ε, τελειώνει ο κύριος ε, Φόξ λέγοντας ότι θέλει να συνεργαστεί με την κυρία Μπερά και τους σκιώδης ηγητές. Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν όλους τους σκιώδης και τώρα... Δεν ξέρω θέλει να επανέλθει η κυρία Μπερά τώρα, να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς να κλείσετε, πώς θέλετε. Πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο για να κάνει την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και την ε, εισηγήτρια κυρία Μπερά για μια πάρα πολύ σημαντική εργασία. Πράγματι πολλή δουλειά έχουμε και χαιρόμαστε που με τις εκθέσεις παίρνουμε πάρα πολύ χρήσιμες ιδέες. Ε, νομίζω ότι ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση του συμβιβασμού ε, ε, ειδικότερα ε, βάσει όλων όσων ακούσα από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα αναφερθώ στα σημεία που ανέφεραν και η συγγήτρια αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν θα αναφερθώ και πάλι στην προαδειοδότηση πριν από τη διάθεση στην αγορά. Νομίζω ότι ήταν σαφή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασιζόμαστε στο φιλο... στη φιλοσοφία του συστήματος αδειοθότησης αλλά και στη μελέτη αντικτύπου την οποία εκπονήσαμε που δείχνει ότι αυτό που προτείνουμε είναι όντω υπέρ τη ασφάλειας και παράλληλα... Ε ακολουθεί τους γρήγορους ρυθμούς ε, εξέλιξης και ε, εισαγωγή στην αγορά των προϊόντων αυτών προς όφελος των πολιτών και προς όφελος βέβαια της καινοτομία στον τομέα αυτό. Όταν ε, μιλάμε για τη διαδικασία παρακολούθησης που προτείνεται στην έκθεση της κυρίας Μπερά, Νομίζω η δική μας διαδικασία, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχο είχε πράγματι την ενίσχυση της ασφάλειας Προτείνουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης που θα δίνει στις αρμόδιες αρχές έγκαιρες πληροφορίες σε σχέση με επικίνδυνα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά, αλλά παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να επιβλέψουμε του, την αξιολόγηση συμβατότητας των προϊόντων αυτών από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Πιστεύουμε ότι πραγματικά ε, σωστά καλύπτουμε τους στόχους αυτούς, όμως βεβαίως ε, μπορούν να γίνουν και βελτιώσεις, γιατί ε, καταλαβαίνω ότι η έκθεση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη της εισηγήτρια αλλά και των υπολείπων ευρωβουλευτών. Τώρα ε, να δούμε ε, κατά πόσο όντω ενισχύει το στόχο που ούτω ή άλλω έχει πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με πολύ χαρά ακούσαμε ότι η συγγήτρια συμφωνεί με την ανάγκη διατήρηση του κανόνα 21. Είναι κάτι το οποίο το είπαμε και χθε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα προϊόντα για τα οποία μιλούμε. Όσον αφορά την. Ε, ε, ε νέα χρήση, την εκ νέου χρήση. Ναι, θα χρειαστεί να το δουλέψουμε αυτό παραπάνω. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η πρόταση της κυρίας ε, Μπερά ε, μπορεί να οδηγήσει σε ε, μια λύση μια συσκευή που προορίζεται για μια χρήση, για παράδειγμα, ίσως να είναι ένα καλό συμβιβασμό. Ευχαρίστως να δούμε αυτή την προσέγγιση που φαίνεται ισορροπημένη και επίση μπορεί να άρει κάποιες νομοθετικές αμφιβολίες σε σχέση με αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Τώρα, όσον αφορά και υπήρχε θέμα μεταξύ των κρατών μελών και για το, ε, στο σημείο αυτό. Είναι όμως μία λεπτομέρεια θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ευρωβουλευτές. Έχουμε δώσει δυνατότητα εξαίρεσης opt-out ε, ακριβώς για αυτό το λόγο. Για τον ορισμό τώρα τον, ε, του αισθητικού σκοπού, ιατροτεχνικά προϊόντα ε, αισθητικής χρήσης. Καταλαβαίνουμε τη, σημασία ενός ορισμού, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι ένα, μια πολύ καινοτόμος και ραγδαία μεταλλασσόμενη αγορά. Μπορούμε να έχουμε έναν ορισμό που να τα καλύπτει όλα. Ε, μπορεί να καταλήξουμε σε μια γκρίζα ζώνη τελικά που μπορεί να συμπεριλαμβάνει κάποιες συσκευές που δεν ε, θα έπρεπε να ρυθμίζονται και δεν καλύπτει άλλες ενώ θα έπρεπε να καλύπτονται. Και σκεφτήκαμε ένα παράδειγμα τα τατουάζ. Και οι μηχανισμοί λοιπόν αναρρόφησης θα εξαιρούνταν. Είναι λογικό αυτό. Όταν είπαμε να υπάρχει θετική λίστα, είναι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους γρήγορους ρυθμούς αυτής της καινοτόμου και ραγδαία μεταλλασσόμενης ε, ε, ε, αγοράς. Όσον αφορά τώρα τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνικά προϊόντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια. Ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη έκθεση για τα δύο θέματα που ε, ετέθησαν. Πρώτον να πω ότι ευχαρίστως να τα εξετάσουμε τη συμπερίληψη ενός ορισμού των γενετικών δοκιμών, των γενετικών ελέγχων Υπάρχει κάτι παρόμοιο και στην έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε και για το πιο οριζόντιο θέμα της υποχρεωτικής ασφάλειας ευθύνης. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ καινοτόμο πρόταση. Να δούμε όμως τις, τεχνικές, τις ε, νομικές πτυχές και να δούμε αν είναι δυνατό από τεχνικής απόψεως ε, βάση των εξουσιών που έχουμε από τις συνθήκες για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Σε γενικές γραμμές χαιρετίζουμε την έκθεση, είναι ισορροπημένη, υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελούν αυτή η βάση βελτιώσεων, ποτέ δεν νομίζαμε ότι είμαστε τέλειοι και είναι και πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα. Η ενίσχυση της παρακολούθησης είναι ένας τρόπος, ε, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αλλά πρέπει να παραμείνουμε και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Καλύψατε πολλά θέματα με τι απαντήσεις σα. Όπως είπαμε είναι περίπλοκη η πρόταση, προκύπτουν διάφορα ω εκ τούτου και ξέρω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε διάφορους τομείς παίρνει διαφορετικό και πορεία από ό,τι εμείς. Εμείς θα πρέπει σαφώς να την ε, δώσουμε σαφή κατεύθυνση της κυρίας Μπερά από την Επιτροπή μας. Ε, όλοι την υποστηρίζουμε σαφώς. Κύριε Μπερά, μήπως θέλετε τώρα να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια είναι τα σχέδιά σας και σε σχέση με το τι γίνεται και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης. Euh, Κύριε Πρόεδρε, ε, σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω. Ζήτησα κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Οι τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 6 Μαΐου στην δική μας Επιτροπή. Η ΕΝΒΗ ψηφίζει τον Ιούλιο στην Επιτροπή. Εμείς, η δική μας ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο, πριν δηλαδή από την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και οι τροπολογίες για την Επιτροπή ΕΝΒΗ πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 13 Μαΐου. Οι τροπολογίες λοιπόν είναι 6 Μαΐου για την ΙΜΚΟ, 13 Μαΐου για την ε, ΕΝΒΗ, Ιούνιος ε, η ψηφοφορία για μας και Ιούλιος για την ΕΝΒΗ με τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Σας απήντησα. Ναι. Αυτά λέει και το δικό μου σημείωμα. Επόμενη λοιπόν ε, συζήτηση θα είναι στις 13 Μαΐου για αυτό το θέμα, έτσι ώστε εσείς και οι σκιώδεις να μπορέσετε να μας παρουσιάσετε τις ε, ε, τροπολογίες και έπειτα να έχουμε κάποιο χρόνο για να εξετάσετε τις συμβιβαστικές, να βρείτε συμβαστικές ώστε να ψηφίσουμε 17 Ιουνίου να έχετε φτιάξει συμβαστικέ και να έχουν όλο το χρόνο να τις μελετήσουν. Έχω μια ερώτηση, λέει η κυρία Παραβάνοβα, για πρακτικούς λόγους. Γιατί 6 Μαΐου είναι η πρώτη ημέρα, είναι η μέρα του Πάσχα, η Δευτέρα του Πάσχα, του Ορθόδοξου Πάσχα και δεν θα είναι πολλοί κόσμος εδώ. Θα ήταν δυνατόν να δεχτείτε την 8η Μαΐου ως προθεσμία γιατί έχουμε αρκετό χρόνο μετά για να εξετάσουμε τις τροπολογίες και η ψηφοφορία θα είναι στα, μέσα, στα τέλη Μαΐου, ε, Ιουνίου και μετά στην έμβη τον Ιούλιο για να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Μήπως μπορούμε λοιπόν αντί 6 Μαΐου να γίνει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 8 ε, 8η Μαΐου. Θα είναι ανακούφιση και για το σύστημά μας. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό το ερώτημα έχει ήδη προκύψει και είχαμε μεγάλη δυσκολία γιατί έχουμε τόση πολλές μεταφράσεις αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να, το, να σας βοηθήσω. Ξέρω πως είναι δύσκολο γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι πράσινη εβδομάδα. Βέβαια μπορείτε να τις καταθέσετε και πριν. Οπότε για την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γιατί πρέπει να ψηφιστούν οι τροπολογίες της κυρίας Μπερά μέχρι τις 18 Ιουνίου ώστε να τις διαβιβάσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ώστε να ληφθεί υπόψη η θέση μας. Υπόψη τους μάλλον. Είναι η τελευταία ημερομηνία για συνεδρίαση της Επιτροπής. Διαφορετικά θα πρέπει να ψηφίσουμε την ίδια εβδομάδα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, οπότε δεν βολεύει. Λυπούμε, αλλά δεν μπορούμε στην πράξη να κάνουμε κάτι. Αν τώρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος καθυστερήσει το δικό της χρονοδιάγραμμα θα το ξαναδούμε. Αλλά το θέμα έχει ξαναπροκύψει, δεν είναι η πρώτη φορά. Είπατε 12 το μεσημέρι για ε, την 6η Μαΐου. Θα ρωτήσω την ε, γραμματεία μου πως τουλάχιστον να γίνει το βράδυ η προθεσμία, 6 το βράδυ τουλάχιστον να έχετε μισή μέρα παραπάνω. Έχει κάποιος κάτι άλλο να πει? Όχι. Κύριε Μπερά, θέλετε να πάρετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το σύνολο των συμμετεχόντων στην Επιτροπή για τις συμβολές τους που ήταν ε, πολύ χρήσιμες. Βεβαίω όλοι έχουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την υγειονομική ασφάλεια για όλους τους ασθενείς στα κράτη-μέλη μας. Ταυτόχρονα κατάλαβα επίσης πολύ καλά ότι μια επιτακτική επιταγή υπάρχει, η επιταγή της καινοτομίας δεδομένη ε, της γρήγορης εξέλιξης ε, αυτού του δυναμικού ε, βιομηχανικού τομέα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας την χαρά μου που διαπίστωσα ότι για τα θέματα διαφάνειας και ανιχνευσιμότητας έχουμε συνένεση μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων καθώς επίσης και η δημιουργία της βάσης δεδομένων που θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό το θέμα διαφάνειας, εποπτείας και παγρύπνησης. Άκουσα τον Κορέα Ντεκάμπος που μίλησε για τη βάση δεδομένων, καθώς και την κυρία Παρβάνοβα για το θέμα των κοινοποιημένων οργανισμών άκουσα τις ανησυχίες σας όσον αφορά το θέμα της εμπειρογνωμοσύνης. Αμφιβο, αμφιβάλλω κατά πόσο μπορούν συστηματικά να προσλαμβάνουν εμπειρογνώμονες οι κοινοποιημένοι οργανισμοί για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θα χρειαστεί να αξιολογήσουν. Και μάλιστα ακόμα περισσότερο γιατί πρότεινα να δημιουργηθεί ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσε κανείς να καλέσει να απαγκαλέσουν μάλιστα οι κατασκευαστές πριν να καταθέσουν ε, τα, ε, τις αιτήσει τους, ώστε το σχέδιο ανάπτυξης τους να είναι σίγουρα ε, αντίστοιχο με αυτό που αναμένεται για τα καινοτόμα προϊόντα όπου δεν υπάρχει αρκετός χρόνος κυκλοφορίας αντίστοιχων και οι εμπειρογνώμονες να μπορούν να επικυρώσουν τα κλινικά στοιχεία που θα δίνουν οι κατασκευαστές έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε την έλλειψη εμπειρογνωμόνων εσωτερικών των κοινοποιημένων οργανισμών. Άκουσα επίσης την ανησυχία της κυρίας Παραβάνοβα ε, όσον αφορά τον ορισμό της απόδοσης, της αποδοτικότητας. Συμφωνώ ε, να προχωρήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό. Έπειτα όλοι μιλήσατε για το θέμα της μιας χρήσης, των προϊόντων μιας χρήσης. Εν γέννη υπάρχει συνένεση να διατηρηθεί το νομικό κενό όσον αφορά το θέμα της ενδεχόμενης επανεπεξεργασίας. Τα προϊόντα μιας χρήσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μία φορά ή αν σε περίπτωση επανεπεξεργασίας μπορούμε να φανταστούμε μια ταξινόμηση εναλλακτική όπως πρότεινα στο κείμενο, δηλαδή υποχρέωση του κατασκευαστή να αποδείξει πως αυτό το προϊόν δεν γίνεται να τύχει εξεργασίες και γιατί. Όσον αφορά τον έλεγχο, συμφωνώ με τον κύριο Κόρε Αντικάμπο, που τόνισε ότι θα πρέπει να γίνονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι, έφοδοι, επιθεωρήσεις στους ε, κατασκευαστές και μόνο από αυτόν τον όρο μπορούμε να εξασφαλίσουμε όντως τη δουλειά μας όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια των πληθυσμών μας. Για να ολοκληρώσω, να πω ότι πιστεύω πως εν γέννη υπάρχει συνένεση για τις διάφο... ανάμεσα στις διάφορες θέσεις ε, των πολιτικών ομάδων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και θα μπορέσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις χωρίς καμία δυσκολία. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας, είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα κείμενο όσο γίνεται πιο ρεαλιστικό, λειτουργικό και εφαρμόσιμο στην πραγματική ζωή. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you, um, very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπερά και όλους τους σκιώδεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που είχαμε αυτή την ευκαιρία για μια πληρέστατη ανταλλαγή απόψεων. Ε, είμαι σίγουρος και το ξέρω ότι θα ε, συνεχίσουν να εργάζονται οι ε, σκιώδεις. κυρία Παρβάνοβα, μας είπατε για την 6η Μαΐου, έχετε μεγάλη πειθό. θα προσπαθήσω να κάνω κάτι, θα είμαστε σε επαφή πάντα και στενή με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί και εκεί θα γίνει πολλή δουλειά, να προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε να στοιχήσουμε τις θέσεις μας. Και θα πάει ή σε δεύτερη ανάγνωση ή στη διαλλαγή, θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και άλλο θέμα. Δεύτερη συζήτηση ε, σήμερα το απόγευμα. Για νέα πρόταση που για πρώτη φορά συζητούμε είναι μια πρόταση οδηγίας εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω ε, το Τζουζέπε Αμπαμόντε που είναι τμήματάρχη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ε, ασφάλειας και εμπιστοσύνη. και τα παλιά μέλη της Επιτροπής μας θα τον θυμούν από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ Τώρα όμως απρόσκοπτα επέρασε σε άλλες θέσεις και άλλα καθήκοντα υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελάτε λοιπόν να μας ε, παρουσιάσετε την πρότασή σας, τη στρατηγική, τις επιλογές μετά από τη μελέτη σκοπιμότητας που κάνατε και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Καλωσορίζω και τον κύριο Γκάστες Γραμμών Σκιώδη ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. κυρία Τούν εκπροσωπεί τον κύριο Σφάμπ, μάλιστα, και εγώ εκπροσωπώ ε, κάποιον άλλον και η κυρία Ρούλε φαντάζομαι ένα δικό της. Α, τον κύριο Έξτρο. Ελπίζω να παραμείνετε για την παρουσίαση. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι... ότι υπάρχει και μία έκθεση ομπρέλα, πώς να την πω, ε, στρατηγικής, μια κοινή ανακοίνωση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, να είναι μεν εύκολη, ανοιχτή η πρόσβαση αλλά και ασφαλής. Ελπίζω λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά, ε, καθώς επίσης και την νομοθετική πρόταση για την οποία έχουμε ορίσει εισηγητή. Χωρί περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζουζέμπε από Μόντε. Έχουμε και τα slides εδώ, τι διαφάνειέ σα μα τι έχετε δώσει και σα δίνω το λόγο με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλου σα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην μακρηγορήσω. 15 λεπτά στόχο βάζω για να μιλήσω κανένα 20 λεπτό με το ΦΠΑ. Ε, η μελέτη αντικτύπου είναι ένας συνδυασμός, συντονισμός μια πολύ μακράς διαδικασίας ε, διαβουλεύσεων ε, για την ασφάλεια στα δίκτυα και στις πληροφορίες μέχρι τώρα. Ήταν εθελούσια η προσέγγιση και βασιζόταν σε συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη ε, και δείτε, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δηλαδή για ασφάλεια ε, των επικοινωνιών. Έχουμε δει λοιπόν ποιες είναι οι διάφορες δυνατότητες και επιλογές στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, ε, για τα κράτη-μέλη. Είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από διάφορους εθνικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο. Για την αντίσταση ε, των συστημάτων αυτών και την ασφάλεια, επίσης συζητήσαμε τη μελέτη αντικτύπου που ε, κάναμε για το EP3R και βεβαίως με τον αρμόδιο οργανισμό μας, την ΕΝΙΣΑ. Κάναμε λοιπόν μια δημόσια διαβούλευση από τις 23 Ιουλίου του 12 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 12 και πήραμε περίπου 180 απαντήσεις. Κυρίως από τη βιομηχανία, από τους ε, ενδιαφερομένους του κλάδου. Επίσης σημειώσαμε και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου Ιδίας Πρωτοβουλίας της 12ης Ιουνίου του 2012 για ε, τις υποδομές επικοινωνιών και το Κοινοβούλιο θυμάστε ότι συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικά μέτρα για καλύτερο συντονισμό των εθνικών κέντρων. Έχουμε ομάδες άμεσης ε, απόκρισης για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όταν υπάρχουν προβλήματα ε, και ε, συμβάντα σε θέματα πληροφορική και τεχνολογίας επικοινωνίας. Επίσης προτείνει το Κοινοβούλιο ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια και την αντοχή ε, των συστημάτων αυτών και να υπάρξει και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινοποίηση παραβίασης ε, της ασφάλειας ε, που αφορά τέτοιου είδους συστήματα. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε στη μελέτη αυτή αντικτύπου. Το πρόβλημα είναι ένα συνολικό, ανεπαρκές συνολικό επίπεδο ασφαλείας στα συστήματα σε σχέση με τα ρίσκα, τις απειλές, τους κινδύνους και τα επεισόδια για τα συμβάντα που επηρεάζουν την ακαιρεότητα και την φερεγγιότητα των συστημάτων. Αυξάνονται όλο και περισσότερο τα περιστατικά, τα συμβάντα, ας πούμε το 2011 οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επιθέσεις αυξήθηκαν παγκοσμίω κατά 81% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έτσι μόνο οι επιθέσεις, όχι όλα τα συμβάντα. Και η περιπλοκότητα των επεισοδίων επίσης αυξάνει. Κάτι άλλο που έχει σημασία 56,8% των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευσή μας είπαν ότι το προηγούμενο έτος είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα σοβαρό συμβάν που απειλούσε ε, τις βασικές υπηρεσίες που οι ίδιοι παρήχαν. Και αυτά τα συμβάντα και επιθέσεις έχουν επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία, σε όλη την οικονομία. Γιατί βασικά στις σύγχρονες κοινωνίες μας και τις ψηφιακές οικονομίες βασιζόμαστε στην τεχνολογία της ε, επικοινωνίας και της πληροφορικής. Δηλαδή όλες οι βασικές λειτουργίες μας που είναι και περίπλοκες βασίζονται στην πληροφορική και επίσης αυτό έχει και ανητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση και την ε, ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γιατί όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, τέτοια επεισόδια, δημιουργείται ε, ένα αίσθημα ανασφάλειας για τις επιγραμμικές υπηρεσίες και σύμφωνα ε, με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο 38% των Ευρωπαίων ανησυχούν και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο, δεν κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές ακριβώς γιατί φοβούνται τέτοιες επιθέσεις ε, και έχουν το ε, αίσθημα αυτό της ανασφάλειας. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τώρα. Το πρώτο, δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ως προς την πρόληψη, ούτε ως προς την απόκρυψη έτσι, στη βορειοδυτική Ευρώπη δεν συγκρίνονται ούτε κατά διάνοια οι δυνατότητες που υπάρχουν σε σχέση με την νότια και νοτιοανατολική ανατολικη Ευρώπη. Και αυτό μας δημιουργεί ένα διπλό πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι, εντάξει, μπορεί να ισχύει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ασφαλείας, διότι ξέρετε ότι κάθε αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος. Αν υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος, ε, κάποιος το αξιοποιεί αυτό, το εκμεταλλεύεται ε, για να επιτεθεί σε όλη την αλυσίδα. Κακόβουλα, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει μια επίθεση σε μια χώρα με χαμηλή αντοχή, αντίσταση και σιγά σιγά να ε, στηθεί ολόκληρη επίθεση κατά χωρών που έχουν και υψηλό επίπεδο προστασίας ε, και αντανακλαστικά. Αυτό είναι το πρώτο ε, σε ό,τι αφορά τις διαφορές. Και η δεύτερη συνέπεια είναι ότι η συνεργασία συνήθως γίνεται ε, μεταξύ μικρού αριθμού κρατών μελών. Και ενώ οι χώρες που υπολείπονται στις δυνατότητές τους εξαιρούνται ή παραγωνίζονται. Δηλαδή γενικότερα η συνεργασία παίζει ρόλο. Ε, συνήθως συνεργάζονται περίπου 10 χώρες μεταξύ τους. Επίσης και έχουν παραθυράκια στους ε, κανονισμούς που ισχύουν και στις νομοθεσίες γιατί η διαχείριση του κινδύνου και των διαφόρων επεισοδίων και συμβάντων στο διαδίκτυο ως προς την ασφάλεια έχουν να κάνουν με εταιρείε τηλεπικοινωνιών και παρόχους γενικότερα ε, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδομών αλλά δεν ισχύουν παντού τα ίδια για όλες τις εταιρείες. Επόμενη διαφάνεια. Δυστυχώς είναι μικρή και δεν ε, φαίνεται πολύ καλά. Προσπάθησα να συνοψίσω τη λογική της παρέμβασης. Το βασικό πρόβλημα είναι η ανεπαρκής ε, προστασία από απειλές προς το δίκτυο. Αυτό προκαλεί ε, κάποιες ε, διακοπές ε, και διαταραχές συνιστά ανασφάλεια για τους πολίτες και απειλή για τη λειτουργία και για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Τι κρύβεται πίσω από το πρόβλημα, είπαμε, έχουμε άνισο επίπεδο δυνατοτήτων και δεν μπορούν να συνεργαστούν όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι μένουν εκτός. Και επίσης Η διαχείριση του κινδύνου δεν είναι ενιαία. Και πολλά από τα συμβάντα και τα επεισόδια δεν τα αναφέρουν καν. Διότι θεωρούν ότι είναι ο σημασίας, δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος, το ρίσκο και δεν τα αναφέρουν καν. Ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι. Στόχος πρώτος, να βεβαιωθούμε ότι οι πάντες έχουν ένα ελάχιστο ε, επίπεδο δυνατοτήτων ή ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας και αντοχής παντού. Δεύτερον, η συνεργασία θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη και όχι τους καλύτερους μαθητές, τους αρίστους. Και ε, η τρίτη ε, προσπάθεια, ο τρίτος στόχος καλύτερα είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η νοοτροπία κουλτούρα ας πούμε, της διαχείρισης του κινδύνου και να αναφέρονται τα σοβαρά συμβάντα και προβλήματα. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε αναλύσει μια σειρά δυνατοτήτων εναλλακτικών. Η πρώτη δυνατότητα είναι αυτή που έχουμε συνήθως business as usual. Τι είχες κάνει, τι είχα πάντα. Να συνεχιστεί η ε, εθελούσια μέθοδος. Το δεύτερο είναι ε, η ε, οδηγία, δηλαδή η κανονιστική προσέγγιση, η ρυθμιστική που αναγκάζει τα κράτη-μέλη να έχουν μια στοιχειώδη δυνατότητα προστασίας ένα ελάχιστο δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη να έχουν μια αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των δικτύων και για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η αρχή αυτή θα πρέπει σε αιτήσια βάση να καταρτίζει στρατηγική και να έχει ένα σχέδιο συνεργασίας με τους υπολείπους για να προλαμβάνονται τα συμβάντα, τα επεισόδια αυτά ή σε περίπτωση που λαμβάνουν χώρα, να αναφέρονται, να ε, συγκρατούνται και να περιορίζονται οι επιπτώσεις. Επίσης, θα πρέπει να είναι ε, σωστή και η χρηματοδότηση και η στελέχωση της αρχής ε, για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων. Το δεύτερο στοιχείο της πρότασης της ρυθμιστικής είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας που να συμπεριλάμβουν και τις 27 χώρες μέλη. Και το τρίτο είναι η επέκταση των απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνου σε μια ε, σειρά υποδομών κρίσιμης σημασίας ε, στις δημόσιες διοικήσεις και η διάδοση επίσης για τα πιο σοβαρά ατυχήματα η ενημέρωση να ε, διαδίδεται σε όλους και να διαβιβάζεται σε όλους τους ενδιαφερομένους. Υπάρχει και η τρίτη λύση που είναι μεικτή, δηλαδή συνδυάζουμε το πρώτο με το δεύτερο, ορισμένα υποχρεωτικά δεσμευτικά μέτρα που να επιβάλλονται στο δημόσιο τομέα ε, και στον ιδιωτικό και να διατηρηθούν και κάποια στοιχεία και κάποια μέτρα σε θελοντική βάση με στόχο να τονωθεί η αναβάθμιση των συστημάτων στα κράτη-μέλη και η συνεργασία επίσης. Επόμενη διαφάνεια. Τι έδειξε η μελέτη, ότι η αμυγός εθελοντική προσέγγιση δεν βοηθάει να φτάσουμε στο στόχο μας. Δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα ε, η αμυγός εθελοντική ε, βάση για διάφορους λόγους, όταν δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Ας πούμε, η αφετηρία Συγγνώμη γιατί μας έφυγε η διαφάνεια. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Yes. Um, uh, the the voluntary approach basically will not will not work because the disparities are too great. Λοιπόν, είπαμε δεν λειτουργεί σωστά η ε, εθελοντική βάση γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές και υπάρχει κίνδυνος να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το χάσμα και αυτό να είναι εις βάρος της σύνολης ασφάλειας στην Ευρώπη και δεν ε, θα μπορέσει να υπάρξει πανευρωπαϊκή συνεργασία. Πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Οι εταιρείε σήμερα, η υπάρχοι κρίσιμων υποδομών, είναι λίγο πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ε, ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια θεωρείται περιττό κόστος και οι εταιρείε δεν καταλαβαίνουν γιατί θα πρέπει να επενδύουν στην προστασία των ε, πληροφοριακών του συστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις άλλες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατανοήσουν αυτό το κίνδυνο και αυτή την απειλή και ε, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει λίγο πιο δεσμευτικό, λίγο πιο υποχρεωτικό και όχι αμυγός εθελοντικό. να υπάρξει δηλαδή μια νοοτροπία, μια κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου και μια επίγνωση του κινδύνου. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η τρίτη επιλογή, η μεικτή προσέγγιση, δίνει μια μερική και μόνο απάντηση στο πρόβλημα χωρίς να επιλύει το πρόβλημα των διαφορών ε, στην προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τη συνεργασία όλων των κρατών μελών. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά αριθμητικά στοιχεία και τι μετρήσαμε, όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία ή τα ε, κοινωνικά ή τις διάφορες ε, επιλογές που έχουμε. Μελετήσαμε επίσης και ε, το επίπεδο ασφαλείας και προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε το κόστος, το διοικητικό και το κόστος της εφαρμογής Είπα ότι θα μιλήσω 20 λεπτά. Δεν έχω πολύ περισσότερο. μιλήσω για το κόστος και μετά θα σταματήσω. Και αν έχετε ερωτήσεις να απαντήσω με χαρά. Επόμενη διαφάνεια. Μεθ' επόμενη μάλλον. Λοιπόν, πρώτον, ποιο είναι το κόστος ε, κατά μέσο όρο και κράτος μέλος. Κατά την άποψή μας δεν είναι και απαγορευτικό. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλες οι χώρες μια αρχή πιστοποίησης ή καταγραφής, ΣΕΡΤ, υπάρχουν ορισμένες που δεν έχουν καθόλου. το κόστος για να δημιουργηθεί αυτή η αρχή εκ του μηδενός είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. το κόστος για την αρμόδια αρχή που θα επιφορτιστεί με τη λειτουργία είναι ένα κόστος της τάξης περίπου των 360.000 ευρώ, αν έχει έξι άτομα προσωπικό. Το πρώτο κόστος στα 2,5 εκατομμύρια είναι άπαξ, ε, το άλλο είναι το κόστος στο μισολογικό και είναι τίσιο, 360.000. Ε, υποθέτουμε ότι όλες οι αρχές θα πρέπει να έχουν την ίδια ιστοσελίδα, ένα κοινό ιστότοπο για να μπορούν να δημοσιεύουν ε, μη ε, ευαίσθητες ε, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα συμβάντα στο διαδίκτυο ε, γενικά όλο αυτό το κόστος για να στηθεί μια ιστοσελίδα είναι 5.000 ευρώ άπαξ, έτσι για, για τη δημιουργία της ιστοσελίδας, συν 2.400 ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση και τη λειτουργία. Ετήσιο κόστος, έτσι ενώ το πρώτο είναι άπαξ. Αυτά, ε, αυτό είναι το κόστος για να στηθεί ε, το σύστημα των δυνατοτήτων και του δυναμικού. Τώρα για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συνεργασίας. Ας ότι εκεί ε, θα συνεδριάζουν τρεις φορές το χρόνο, ας πούμε, έτσι, σε πραγματικές συνεδριάσεις, στον ίδιο χώρο. Εκεί το κόστος ανακράτος μέλους θα είναι περίπου 6.000 ευρώ, έχουμε υπολογίσει. Είναι το κόστος για να μεταβαίνουν οι αρμόδιες στις συνεδριάσεις. Α, κάτι άλλο που είναι σημαντικό και πρέπει να σας πω, είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν και να αποδείξουν ε, την ετοιμότητά τους να συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκές ασκήσεις. Ο ΕΝΙΣΑ το 2010 έκανε μια τέτοια προσωμείωση, έκανε μια τέτοια άσκηση και πιστεύουμε ότι για να συμμετέχουν όλοι και τα 27 κρατημέλη, αυτό θα έχει ένα κόστος περίπου 55.000 ευρώ. Το χρόνο Ας πούμε αν υπάρχει μια άσκηση κάθε χρόνο. Κάτι άλλο επίσης που έχει σημασία είναι ότι στο μηχανισμό συνεργασίας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, μοιράζονται ευαίσθητες προφορίες και προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ασφαλή υποδομή αν θα πρέπει να στηθεί η υποδομή αυτή από το 0 και πάλι, το κόστος είναι περίπου 10.000 ευρώ. Όχι, 10 εκατομμύρια διορθώνει ο μιλητής. 10 εκατομμύρια ευρώ, που είναι αυτό που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εταιρεία Orange για να έχει ε, τα κυκλώματα αυτά ε, και το, τον ιστότοπο που χρειάζεται. Εάν αποφασίζουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, η φυστάμενη υποδομή όπως είναι το s το κόστος είναι μικρότερο βεβαίως είναι κόστος προσαρμογής και φτάνει περίπου στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πάλι αυτό εφάπαξ καταβάλλεται στην αρχή. Το επόμενο slide. Προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε εδώ όσο καλύτερα μπορούσαμε ήταν και πάρα πολύ δύσκολο και πάλι αυτό, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτά τα δεδομένα. Το κόστος για τον ιδιωτικό τομέα και για τις δημόσιες διοικήσεις. Ιδού λοιπόν σε αυτό το πίνακα ποιο είναι το κόστος διαχείρισης του κινδύνου και ε, δημιουργίας λύσεων ασφαλείας ε, που να αναλογούν ε, στην σοβαρότητα των κινδύνων που έχουμε εντοπίσει και ανιχνεύσει. Υπολογίσαμε λοιπόν ότι κατά μέσο όρο το κόστος Α, συγγνώμη, παρένθεση. Το συνολικό κόστος είναι περίπου της τάξεως του ενός εκατομμυρίου μέχρι 1,9 εκατομμύριο. Αυτό πώς έχει υπολογιστεί. Α, διορθώνει ο μιλητής. Όχι εκατομμύριο, δισεκατομμύριο. Τα βλέξα λίγο εδώ με, με το pointer δισεκατομμύρια. ένα με 1,9 δισεκατομμύρια. Και αυτό έχει υπολογιστεί για όλες τις εταιρείες και για όλες τις δημόσιες διοικήσεις ε, που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα κόστος στόχο που είναι βέλτιση στις πρακτικές του κλάδου αν πάνε όλα καλά δηλαδή, ε, μια μελέτη που έκανε η Ραντ, η ενέργεια έχει παραδοσιακά τις καλύτερες επιδόσεις στη διαχείριση κινδύνου. 6,6% λοιπόν δίνουν οι εταιρείε ε, ενέργειας από το προπολογισμό ε, της ε, επικοινωνίας και της πληροφορικής για ασφάλεια. 6,6%. Γιατί οι περισσότεροι είναι ελεγκτές των δεδομένων. Κάναμε λοιπόν δύο κουρέματα, όπως τα λέμε, στο θεωρητικό μέγιστο κόστο. Το πρώτο κούρεμα 40% και το δεύτερο 70% ακόμα μεγαλύτερο και καταλήξαμε σε αυτά τα στοιχεία. Συνολικά το κόστος Αυτοί που διαχειρίζονται λοιπόν κρίσιμες υποδομές όπως και οι δημόσιες διοικήσεις θα έχουν ένα κόστος συνολικά, είπαμε, ε, ε, ανάμεσα σε 1 και 1,9 δισεκατομμύρια. Αυτή η πρόταση αφορά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές εξαιρούνται και για τις μικρομεσαίες το κόστος είναι 2.500 με 5.000 ευρώ ανά εταιρεία. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό και δεν και πολύ μεγάλο κόστος. Αν δει κανείς πόσο κοστίζει ένα επεισόδιο ηλεκτρονικό που διαταράσει την ασφάλεια. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, είδαμε μια τέτοια κατάσταση, έγινε μια μελέτη από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το κόστος για μια μικρή εταιρεία, αν υπάρχει ένα επεισόδιο στην ασφάλεια, είναι 15 ε, με 30 χιλιάδες ευρώ. Για μικρή εταιρεία έτσι και για μεγάλη εταιρεία δεκαπλασιάζεται. Και τέλος, ε, έρχομαι στην τελευταία διαφάνεια. Ποιο είναι το μέσο κόστος για κάθε κοινοποίηση ε, προβλήματος ασφαλείας. είναι μελιτέο, είναι ένα κόστος ενός email περίπου. 125 ευρώ. 10 με 20% των κοινοποιήσεων ακολουθούνται από έρευνα. Δίνεται συνέχεια δηλαδή. Και έχουμε αξιολογήσει το μέγιστο κόστος για να, ε, αν χρειαστεί, οι εταιρείε να παρακολουθήσουν, να δώσουν συνέχεια με έρευνα. Τότε το μέγιστο κόστος είναι 25.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε την πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ίσως να έχουμε μια μεικτή προσέγγιση. Αυτό είναι καλύτερο. Όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε υποθέτω ότι και οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου. Είναι και εδώ η κυρία Γκέπχαρτ, πρώτα όμω η κυρία Τούρνεν. Και ο κύριο Καρθέ Ραμών αν θέλει να πάρει το λόγο. Όποιος θέλει το λόγο, ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαμπ δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε μου ζήτησε να σας διαβάσω ουσιαστικά το κείμενο το οποίο παρουσίασε. Ήθελε εκείνος να σας το διαβάσει, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ. Θα ήθελα καταρχάς να πει ότι χαίρεται όλος ιδιαιτέρως ε, που η δουλειά για την, ασφαλεία, για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών, όπως επίσης και για τη στρατηγική περιασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αρχίζει επιτέλους σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί όλο και περισσότερο υπάρχουν ε, επιθέσεις στο διαδίκτυο και γι' αυτό επικροτεί τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελε να υπενθυμίσει κάποιες, ε, κάποια βασικά περιστατικά που δείχνουν πόσο, πόσο κοντά είναι ε, σε κάθε ένα από εμά και πόσο ευάλωτοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο που όλο και περισσότερο ψηφιοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, κοινωνίες. Τρία παραδείγματα. Το 2007 επιθέσεις hackers κατάφεραν να παραλύσουν σχεδόν μια ολόκληρη χώρα, την Εστονία, και, δημοτικοί, και δημόσιοι φορείς ε, ενεπλήγησαν πάρα πολύ. Το 2011 το Sony PlayStation ε, ε, ήταν ετυχήμενο επίθεσης, κλάπησαν πάρα πολλά στοιχεία, θα θυμάστε. Και αυτό το μήνα ένα σύστημα θέρμανσης ε, στη Γερμανία φάνηκε πόσο ευάλωτο ήταν. Τόσο ευάλωτα είναι που μπορούν πολύ εύκολα, μπορεί κανείς να τα σβήσει, να σβήσει το σύστημα θέρμανσης μέσω ίντερνετ. Για να δούμε ακριβώς πόσο μεγάλο, πόσο ευάλωτοι είμαστε, θα έπρεπε κάθε ε, καταναλωτής να ζητήσει από την Επιτροπή να πάει σπίτι του να διορθώσει το πρόβλημα να δει πόσο ευάλωτος είναι κανείς. Καθένας από μας μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ από έλλειψη ασφάλειας το ίμιση των κρατών μελών μόνο έχουν μια εθνική στρατηγική ασφάλεια ε, στον χώρο, οπότε μια κοινή προσέγγιση είναι όλο και πιο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της ε, ρύθμισης και της ευελιξίας σε ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο όλο και συνεχώς αλλάζει και επίσης συνεχώς εξελίσσεται. Επομένως ο εισηγητής θα ήθελε να ε, με επί τη της σημερινής κοινή συζήτηση να λάβει κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που του φαίνονται σημαντικά και τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να απαντηθούν στις ε, επικείμενες νομοθετικές διαδικασίες για το διαδίκτυο, για την ε, ασφάλεια για την οδηγία που αφορά την ασφάλεια των δικτύων και της, των πληροφοριών. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ μιας κουλτούρας ε, ανάληψης, εξορρόγησης κινδύνου του κλάδου, η οποία όμως όμως δεν σημαίνει μια, έναν κατάλογο συμβατότητας που να είναι πάρα πολύ βαρύς, ε, Δηλαδή δεν σημαίνει ότι απλώς επειδή κάποιος έχει καλύψει όλα τα στοιχεία συμβατότητας ότι έχει ε, ε, καθαρίσει. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, προβλήματα γύρω από την αξιολόγηση κινδύνου. Μιλήσατε πολύ για το κόστος. Πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα τους πίνακες που μας παρουσιάσατε. Δεν μπόρεσα να τους διαβάσω γιατί ήταν πάρα πολύ μικροί. Δεν ακούσαμε από εσά επαρκεί για το πώς καταλήξατε στα νούμερα αυτά. Και αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο κύριο Φαμπ. Και το λέω αυτό γιατί είχα πολύ κακή εμπειρία και στο παρελθόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με εκτίμηση κόστους. Οπότε ελπίζω τέλος πάντων να το έχετε διερευνήσει επαρκώς και είμαι σίγουρη ότι και ο κύριος Φαμπ θα ήθελε να μάθει πώς καταλήξετε σε αυτά τα νούμερα. Το ερώτημα που έχει να θέσει είναι, λέτε ότι είναι πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να υπάρξει μια κοινή ε, προσέγγιση ε, κρατών μελών και ευρωπαϊκού επίπεδου. Ο εισηγητής θα ήθελε λοιπόν να μάθει περισσότερα σε σχέση με τις ιδέες που υπάρχουν για ένα κοινό ε, εργαλείο ασφάλειας γιατί έχουμε κάποιες οδυνηρές εμπειρίες IT εργαλείων που η διαχείριση τους γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το σύστημα για τις θεωρήσεις και το σύστημα Σέγγεν. δεν συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο συνεργασίας ε, οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς. Δεν έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση, η ΕΝΙΣΑ, η Europol, η Eurojust, ε, ε, όλοι αυτοί οι φορείς να συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο συνεργασίας. Ο Ανδρέας Φάμπ είχε επίσης ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. το βασικό εργαλείο είναι η στρατηγική ασφάλεια στο κυβερνοχώρο. Ο εισηγητής Χαίρεται που έχουν καλυφθεί ορισμένα σημαντικά στοιχεία, όμως κάποια από τα στοιχεία της Επιτροπής φαίνονται κατά τη αδύναμα. Αναφερθήκατε μόνο στη δημόσια διαβούλευση της περασμένης χρονιάς 160 απαντήσει πήραμε μόνο. Δεν είναι και κανένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Μιλήσαμε πάρα πολλέ φορέ εδώ ε, για τη δημόσια διαβούλευση και συνήθω είναι πάρα πολύ συχνά τόσο λίγες οι απαιτήσει γιατί δεν χρησιμοποιεί όλε τι επίσημε γλώσσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτέ οι 160 απαντήσει επαρκούν για να δικαιολογήσουν την προσέγγιση που επιλέξατε. Κάτι ακόμη που ενδιαφέρει τον εισηγητή πώς έχετε ε, σκοπό να εξασφαλίσετε τα ε, ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα όταν υπάρχουν επιθέσεις, για παράδειγμα, στον κυβέρνοχώρο. Και τέλος, Όσον αφορά το διάλογο με τις τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την εστίαση σε εταίρους ε, που έχουν παρόμοια άποψη με τη δική μας. Όμως ε, πολλές ε, κυβερνοαπειλές προέρχονται από χώρες που προφανώς δεν έχουν την ίδια άποψη μαζί μας και πώς έχετε σκοπό να το αντιμετωπίσετε αυτό. Ο εισηγητής θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι περιμένει με αγωνία τις επόμενες ε, συνεδριάσεις και συζητήσεις με τους συναδέλφους ε, και άλλους φορείς. Και τώρα να σας πω για το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα 25 Απριλίου έγινε η μελέτη, η ε, παρουσίαση της μελέτης, ακρόαση 18 Ιουνίου Σχέδιο γνωμοδότησης πρέπει να είναι έτοιμο στις 20 Ιουνίου για μετάφραση. Αυτά. Α, και για το σχέδιο ψηφίσματος. Για τη στρατηγική ασφαλείας. 25 Απριλίου σήμερα έγινε η παρουσίαση, εξέταση του σχεδίου 7 Μαΐου και προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 27 Μαΐου, εξέταση των τροπολογίων 18 Ιουνίου και θα έπρεπε κανονικά να το ψηφίσουμε εδώ ε, στις 8 ή 9 Ιουλίου για να πάει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Αυτά για το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. thank you. Uh, and thank you. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Σφάμπ για τη δουλειά του. Ελπίζω να υπάρξουν απαντήσεις στα ερωτήματά του. Ο κύριος Γκαρσές Ραμόν. Θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα? Μετά δεν ξέρω και η κυρία Ρούλε μπορεί να θέλει να πάρει το λόγο και εγώ βέβαια μετά γιατί και εγώ είμαι σκιώδης συζητητής. Κύριε Γαρσές Ραμόν πρώτα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος σε αυτή την πρώτη μου τοποθέτηση διότι μπαίνουμε στην πρώτη φάση των κοινοβουλευτικών εργασιών για ένα θέμα με τεράστια περιπλοκότητα, όπως φάνηκε άλλωστε από την παρουσίαση αλλά και τα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας. Θα χρειαστεί λοιπόν μεγάλη προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις στα προβλήματα ε, τα οποία τίθενται. Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχούν ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή δύο πράγματα. Και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, με την προλαλήσαντα, συγγνώμη. Ε, σε δύο θέματα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, θα απαντηθούν στη συνέχεια. Ε, και ποια είναι αυτά. Πώς θα οριστεί η σχέση, η επικοινωνία μεταξύ αυτής της οδηγίας που συζητούμε εδώ και της οδηγίας για θέματα ασφάλειας στον κυβερνό χώρο που δεν είναι η ίδια οδηγία προφανώς, αλλά έχουν κάποια συνάφεια μεταξύ τους. Ε, πολύ στενή. Θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, βλέπει αυτή τη διασύνθεση εκεί. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση, το πρώτο μέλημα και ένα δεύτερο. σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, των πολιτών εν γέννη. Το δικαίωμα φέρει πίν στην πρόσβαση και τη χρήση των δικτύων, αλλά με εγγύησει. Όχι μόνο ασφαλιστικές δικλίδες, που σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας, αλλά ε, και ως προς τα δικαιώματα της απρόσκοπτης πρόσβασης, όχι χωρίς περιορισμό η περιστολή ελευθεριών ή θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην έκφρασή τους μέσα από τις νέες τεχνολογίες ε, της ε, επικοινωνίας, της πληροφορίας και των δικτύων. Γιατί είναι όλη αυτή μια νέα πραγματικότητα. Και ένα τρίτο είναι το οικονομικό πεδίο. Το ακούσαμε και από την προηγούμενη ομιλήτρια. Κοιτάζω εδώ πέρα τους αριθμούς που μας δίνετε και θέλω να ρωτήσω, καλά πότε έγινε αυτή η οικονομική μελέτη, χρονικά, ημερομηνία, ποια περίοδο εννοώ, πότε τα υπολογίσατε όλα αυτά. Και πώς καταλήξετε σε αυτά τα συγκεκριμένα νούμερα. Από τη μια ε, ε, μιλάτε για ένα με δύο λέει δις. Είναι μεγάλη διαφορά. Ή 1.500 ε, με 5.000 ή 2.500 με 5.000 ευρώ. Κάθε φορά είναι το διπλάσιο από το προηγούμενο. Χωρίς να μπω βέβαια σε λεπτομέρειες, θέλω να ρωτήσω πότε ακριβώς έγινε αυτή η οικονομική μελέτη και πώς υπολογίσατε αυτά τα ποσά. Και τέλος, κάνατε καμιά μελέτη, ανάλυση, πρόβλεψη για το πώς έχουν οι σχέσεις ανάμεσα στις δημόσιες επενδύσεις για να είναι συγκεκριμένη και αποτελεσματική στην πράξη αυτή η μελέτη. Τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά και τι επιπτώσεις θα έχει γενικότερα. Εκ των υστέρων. Ε, στις δημόσιες υπηρεσίες. Ε, το έχετε σκεφτεί αυτό για τις δημόσιες επενδύσεις ρωτώ σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις και τι συμφέρον θα έχει το δημόσιο και τι συμφέρον ο ιδιώτης. Αυτά προς το παρόν, κάποιες πρώτες σκέψεις. Γνωρίζω ότι εντός του χρόνου διαγράμματος που έχουμε ορίσει υπάρχει ανάγκη να συναντηθούμε ξανά και να ανταλλάξουμε απόψεις πιο εμπεριστατωμένες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πολύτιμα σχόλια. Κυρία Ρούλε, θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω κι εγώ τη συζήτηση ε, λέγοντας ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του κυρίου Γκαρσέ Σεραμών ε, σε σχέση με ορισμένα ζητήματα. Η επιλογή των μέσων που κάνατε Νομίζω ότι στο πλαίσιο των ευρύτερων ε, προγραμμάτων, ε, των εθνικών προγραμμάτων συνεργασίας, ε, ομάδων εκτάκτου, ανάγκης, νομίζω ότι δεν είναι σαφές αν χρειάζεται ένα νομικό μέσο ή όχι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η λογική. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, επιμείνατε μάλλον ε, σε όλες αυτές τις ε, απαιτήσει για κάτι που σε μένα φαίνεται ότι είναι ε, ευρύ φάσμα οργανισμών στο άρθρο 14, ας πούμε λέει ότι οι δημόσιε διοικήσεις και οι φορείς της αγοράς πρέπει να, μπαίνουν, να παίρνουν τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν συστήματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ευρύ για να μπορέσει να το εφαρμόσει ένα κράτος μέλος. Και μου φαίνεται ότι είναι και αόριστο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, αλλά νομίζω ότι η διαχείριση του κινδύνου είναι πάρα πολύ ευρύ πράγμα και αν θέλετε πραγματικά να επιβάλλετε τις διατάξεις αυτές και να ζητήσετε από όλους τους φορείς της αγοράς ε, αλλά ε, και τις ε, δημόσιες διοικήσεις να, το, να εφαρμόσουν αυτό το πράγμα που ζητάτε, πραγματικά αυτό είναι κάτι που επιβάλλει πολύ ουσιαστικό και μεγάλο διοικητικό κόστος. και νομίζω ότι η εκτίμηση του κόστους που κάνατε για την εφαρμογή και την επιβολή κυρώσεων ε, συνάδει με αυτά που μας είπατε. Είπατε ένα δις ε, σε όλη την Ευρώπη, τέλος πάντων ένα τομέα, δεν κατάλαβα ακριβώ πώς το είπατε. Αυτό τέλος πάντων το κόστος συμμόρφωσης ε, το αναφέρατε, αλλά μιλήσατε για κόστος επιβολής και δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι πρακτικό κάτι τέτοιο γιατί δεν είναι ένα πολύ επιλεκτικό μέσο και το, να αντιμετωπίζουμε πραγματικά προβλήματα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρούμε. Για παράδειγμα, ο εξοπλισμός. Πρέπει όλος ο εξοπλισμός που παρέχεται να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Και μιλάω και για το λογισμικό. Ε, να υπάρχουν κάποια μέτρα στον κυβερνοχώρο και μιλάω για την τεχνολογία. Είπατε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποια εθελοντικά μέτρα σε σχέση με ε, την εκπαίδευση γύρω από τα θέματα αυτά. Μπορεί αυτά να είναι πιο εφικτά σε αυτό το τομέα από ότι, ε, από για μια οδηγία την οποία όμως προσεγγίζεται με πάρα πολύ αόριστους όρους. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν κάθε δυνατότητα διερεύνησης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ναι, αλλά τι κόστο μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε πόσοι άνθρωποι πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί για να το κάνουν αυτό το πράγμα, να πηγαίνουν να επιθεωρούν κάθε επιχείρηση, κάθε μεγέθου, ε, ε, για να βεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τα κριτήρια, με τι προδιαγραφέ. Τι να σα πω, δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιο ότι δεδομένος δεδομένης της και της τάση μείωση των δημοσίων δαπανών, ότι κάτι τέτοιο θα ειδωθεί πάρα πολύ ευνοϊκά από τα κράτη-μέλη, εκτό αν εσείς έχετε κάτι άλλο υπόψη σας και μπορείτε να με καθησυχάσετε. Θέλουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν, αλλά υπάρχουν κάποιε ανησυχίε. Και για τη στρατηγική. Κοιτάξτε, αυτή η στρατηγική πτυχή είναι το θέμα που με ανησυχεί περισσότερο και Έχουμε και εμεί ένα τμήμα αξιολόγηση αντικτύπου και μια σχετική αξιολόγηση. Βλέπω ότι ο συνάδελφο είναι εδώ, μάλιστα, ή συνάδελφο, είπε το ίδιο πράγμα. Έκανε και εκείνη μια αξιολόγηση τη δική σα αξιολόγηση και είπε ότι παραθέτω λόγω του ότι πρέπει να καταδειχθεί αναλογικότητα του προτινόμενου μέτρου, πρέπει να γίνει μια πραγματική αξιολόγηση του κόστους ε, ε, της επιβολής του μέτρου αυτού, όπως επίσης και το επίπεδο λεπτομέρειας, το επίπεδο άχθος που θα σήμαινε αυτό για τους φορείς ε, και κατά πόσο όντως κάτι τέτοιο θα ε, ε, χρήζει όντως τόσο λεπτομερούς ρύθμισης. Δηλαδή, Εγώ ε, το κατάλαβα καλά ή έχετε τίποτε άλλα ε, πάρα πολύ ε, αποστομωτικά επιχειρήματα να μου παραθέσετε για να μου εξηγήσετε αν το κατάλαβα καλά ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω με τη σειρά στα σχόλια αυτά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον υπολογισμό του κόστους. Βασιστήκαμε σε στοιχεία της Eurostat και σε στοιχεία ιδιωτικής ανάλυσης. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι πρόκειται για έναν αναδυόμενο τομέα, οπότε τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να τα βρει κανείς. Η αξιολόγηση λοιπόν αντικτύπου έγινε πέρυσι και χρησιμοποίησαμε τα, τα πιο πρόσφατα και τα καλύτερα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Όταν δεν υπήρχαν στοιχεία, έπρεπε να σκεφτούμε θεωρητικά μέγιστα από νούμερα και μετά να κάνουμε εκτιμήσεις. Σε αυτό το τομέα δεν είναι σπάνιο κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη μελέτη της Price Waterhouse, όταν βλέπουν το, εξετάζουν το κίνδυνο ρήξης της παραβίασης της ασφάλειας, δίνουν ένα φάσμα 15 με 30 χιλιάδες ας πούμε. έχει, ε, το Εθνικό, ο Εθνικός Οργανισμός έχει εκτιμήσει το κόστος του κυβέρνου εγκλήματος μέχρι ε, ανάμεσα στις 20 και στις 50.000 λίρες. Δεν υπάρχουν στοιχεία, οπότε δεν είναι ασυνήθιστο και μάλλον είναι συντηρητικά τα νούμερα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να σκεφτούμε ένα μέγιστο αυξητικό κόστος που μπορεί να προκληθεί λόγω των νέων νομοθετικών απαιτήσεων. Όλος ιδιαιτέρως ρωτήσατε κυρία Τούν πώς υπολογίσαμε το κόστος, γιατί δεν μπορούσατε να το δείτε. Για τους προμηθευτές, τους παρόχους κρίσιμων υποδομών και τους ε, διαχειριστές. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να υπολογίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στον στόχο δαπάνης ε, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές. Οπότε αυτό το ιδανικό επίπεδο είναι 6,6% του προϋπολογισμού IT μιας εταιρείας. και προσπαθήσαμε να βάλουμε αυτό στις ε, πραγματικές δαπάνες των διαφόρων ε, ε, τομέων. Οπότε το επίπεδο στόχος προσαρμοζόταν με την φυσική αύξηση των δαπανών, γιατί υποθέτει κανείς ότι δεν είναι κάτι στατικό διαχρονικά, αλλά που θα αυξάνεται γιατί θα είναι τα περιστατικά πιο συχνά και πιο περίπλοκα. Και αυτό ήδη δείχνει πόσο συντηρητικοί ήμασταν στον υπολογισμό του κόστους. Το συνολικό λοιπόν ανώτατο θεωρητικό ποσό είναι 3 δις ευρώ για τις 42.500 εταιρείες και διοικήσεις που θα επηρεαστούν από τις απαιτήσει αλλά αυτό θα πρέπει να μειωθεί από το κούρεμα που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι όλες αυτές οι εταιρείε, ας πούμε, μια τράπεζα είναι ελεγκτή στοιχείων. Ήδη τώρα υποχρεούται ε, σε, κάποιο βαθμό να θεσπίσει ασφα... Ε, προδιαγραφές ασφάλειας λόγω του πλαισίου για την προστασία των δεδομένων. Θα υπάρξουν κάποιες επιπλέον δαπάνες που θα πορέουν από τη δική μας ε, πρόταση που θα πρέπει να φτιάξουν, αλλά γι' αυτό και έχουμε αυτό το, φάσμα. Πρέπει να είμαστε λίγο εφάνταστοι εδώ, αλλά πιστεύουμε πως αυτά τα νούμερα μπορούν να σταθούν. Και πάλι, επαναλαμβάνω, πολύ συντηρητικά τα έχουμε υπολογίσει. Τώρα, η σχέση μεταξύ αυτής της ε, οδηγίας και της οδηγίας περί κυβερνοεγκλήματος που αναφέρατε. Ενημέρωση, βοήθεια στις υποδομές. Η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις οδηγίες, κατά τη γνώμη μου, Μάλλον, η οδηγία για το κυβερνοέγκλημα είναι οδηγία περί ποινικού δικαίου. Ποινικοποιεί και εισάγει κοινού ορισμούς του κυβερνοεγκλήματος και των κυβερνοεπιθέσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κάνουμε εμείς, εμείς ασχολούμαστε όχι με το κυβερνοέγκλημα, δεν μας απασχολεί το ε, ο ποινικό χαρακτηρισμός μιας επίθεσης. Εμείς ασχολούμαστε με τη βελτίωση του δικτύου μέσω μιας καλύτερης προετοιμασίας, δηλαδή την θέσπιση προληπτικών μέτρων και των καλύτερων μέτρων ανταπόκριση σε τέτοιες επιθέσεις. Περισσότερο δηλαδή ασχολούμαστε, αν θέλετε, με τα πολιτικής φύσης μέτρα που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να αναχαιτήσουν τις επιθέσεις και τον αντίκτυπό του στην οικονομία και στην κοινωνία. Εσείς αναφέρατε πώς, μπορούμε να, πώς μάλλον εξισορροπήσαμε το κίνδυνο διαχείρισης, δηλαδή την εισαγωγή ή την ε, μιας ε, νοοτροπίας διαχείρισης κινδύνου με τα συγκεκριμένα μέτρα. Ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η στρατηγική κυβερνοασφάλειας παρέχει μια σειρά μέτρων που είναι βασικά για αυτή την οδηγία. Ιδιαίτερα μόλις ξεκινήσαμε μια, ένα, ένα, δηλαδή μια βάση ε, ε, ασφάλειας δικτύου που θα είναι μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ώστε να εντοπιστούν οι πρακτικές και τα κίνητρα που στόχο θα έχουν να εθαρρύνουν ε, τους παρόχους των υποδομών αυτών να προβούν και να χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες πρακτικές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι στον τομέα αυτό δεν υπάρχει ε, η μαγική λύση και η οδηγία δεν ορίζει το είδος των ε, λύσεων ασφαλείας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διότι σε αυτό συμφωνώ, κυρία Τούν, μαζί σας, ότι κάτι τέτοιο θα έδινε θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας ε, απαρίθμησης ε, λύσεων και καλύτερα είναι κανείς να μπορεί να εντοπίσει τους κινδύνους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και να φτιάχνει μέτρα που να είναι αντίστοιχα και αναλογικά του κινδύνου. Να θεσπίσει δηλαδή μέτρα ασφαλείας που βασικά να αντικατοπτρίζουν και να είναι ανάλογα και με τη σοβαρότητα του κινδύνου που, που έχει εντοπιστεί κάθε φορά. Είπατε ότι μέσα στο μηχανισμό συνεργασίας τα κράτη-μέλη μοιράζονται ε, πληροφορίες και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένταση ανάμεσα στην απέτηση της ε, διαβίβασης πληροφοριών και της προστασίας των δεδομένων. Σας παραπέμπω στο εκτιμώντας 39 της πρότασης που λέει ότι η διαβίβαση πληροφοριών θα είναι απαραίτητη, είναι απαραίτητη ώστε να συμμορφωθεί κανείς με τις νομικές ε, απαιτήσεις. Είναι απαραίτητο δηλαδή να ανταποκριθούμε στους στόχους ε, δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκει αυτή η στόχη και ως τέτοιο είναι θεμητό και εντάσσεται στο σχετικό άρθρο της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων. Τώρα ένα σημείο που συνδέεται περισσότερο με το στρατηγική της οδηγίας. Το γεγονός ότι οι απειλές προέρχονται από χώρες που δεν, σέβονται, δεν σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο, όπως είπατε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και όλα τα μέτρα στην οδηγία ισχύουν για κάθε είδους επίθεση. Δηλαδή άσχετα με το ποια θα είναι η φύση της επίθεσης, είτε είναι φυσική καταστροφή λόγω πλημμύρας, είτε πρόκειται για ανθρώπινο λάθος στην ε, συντήρηση του ε, δικτύου, είτε αν είναι ε, κυβερνοέγκλημα ή κυβερνοκατασκοπία που προέρχεται από το εξωτερικό, η οδηγία ισχύει λοιπόν για κάθε είδους περιστατικό που μπορεί να συμβεί στην Ένωση άσχετα από την προέλευση του, του περιστατικού. Και έπειτα οι πολύ σωστές παρατηρήσεις ε, του Προέδρου. Γιατί χρειαζόμαστε τον τρίτο πυλώνα που είναι οι απαιτήσει ασφαλείας που θα πρέπει να εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα και στι δημόσιε διοικήσει και το κόστος. Πιστεύουμε πως χωρίς τον τρίτο πυλώνα όλος αυτός ο χάρτινος πύργος μπορεί να καταρρεύσει. Και γιατί αυτό... Καταρχήν, διότι είναι απαραίτητο να έχει κανείς ε, καλή συνεργασία και σύμπραξη ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, γιατί ο ιδιωτικό τομέα κατέχει τις υποδομές. Το διαδίκτυο δεν το διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις, αλλά ο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα επίσης εν γέννη είναι πολύ απρόθυμος να μοιραστεί με οποιονδήποτε τέτοιου είδους πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της μελέτης αντικτύπους, ότι δηλαδή τα περισσότερα περιστατικά δεν αναφέρονται και δεν τα παρατηρεί και κανείς, γιατί υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό περιστατικών που παίρνουν δημοσιότητα. Και αυτό όταν είναι πολύ αργά πια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφοράς για δύο λόγους. Καταρχήν, διότι η, ε, τέτοιου είδους απαιτήσεις αναφοράς διευκολύνουν την αρχή ασφάλειας να προετοιμάσει μια πιο αξιόπιστη στρατηγική, αν θέλετε. Και επίσης πιο ε, αξιόπιστη συνεργασία ως απάντηση, που είναι πολύ σημαντική. Ε, δεύτερο είναι ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια ε, υποχρέωση για την ε, εταιρεία γιατί έτσι οι εταιρείε πιστεύουμε θα προσέχουν περισσότερο στη διαχείριση του κινδύνου που εντοπίζουν. Δεν θα είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται όλα τα περιστατικά, μόνο τα σοβαρότερα τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές οι εταιρείε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στον τομέα της ε, τηλεπικοινωνίας, όπου έχουμε την ίδια απέτηση ακριβώς, Μέχρι στιγμής ο αριθμός των περιστατικών που έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη την Ένωση είναι μόνο 61. Μόνο 61 περιστατικά έχουν ε, κοινοποιηθεί. Αναμένουν βέβαια ότι διάφορα περιστατικά που αφορούν ε, όλη αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που θα έχει αυτή ροτεριστεί περισσότερο, ε, ο αριθμός των περιστατικών θα αυξηθεί. Αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να κοινοποιούνται όλα τα περιστατικά που εντοπίζονται. Τώρα, ε, και πάλι, όλα αυτά θα δείτε στο μελέτη αντικτύπου. Επί τη βάση των συστάσεων και των εκτιμήσεων της ΕΝΙΣΑ, μόνο το 10% όλων των κοινοποιήσεων που πάλι θα εμπίπτουν σε κάποιο φάσμα, θα πρέπει να ακολουθηθούν από συγκεκριμένη έρευνα, ανάλογα με το μέγεθός τους έχουμε δώσει στοιχεία. Μπορέσα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην μελέτη αντικτύπου τέλος. Τέλος, η αξιολόγηση που κάνουμε τώρα όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου εδώ στην Ευρώπη δεν βοηθάει πολύ, ούτε μας καθησυχάζει ιδιαίτερα, διότι γνωρίζουμε θα σας πω κάτι που προέκυψε σαφέστατα από την δημόσια διαβούλευση. 31% των απαντώντων δεν έχουν καμία διαδικασία για να διαχειριστούν τον κίνδυνο. Και το 54% και όλε αυτέ οι εταιρείε, αν φανταστείτε, είναι εταιρείε που είναι πολύ ξεκιωμένες με τα θέματα αυτά, γιατί είναι εταιρείε που ασχολούνται με την ασφάλεια και δεν έχουν καν προπολογισμό αφιερωμένο στην, στην ασφάλεια του δικτύου. Χρειάζεται λοιπόν, πιστεύουμε πως χρειάζεται οπωσδήποτε οπωσδήποτε να προωθήσουμε ε, αυτήν την ε, οδηγία. Κάτι ακόμα που είπε η κυρία Τούν για τη συμμετοχή της Europol και της Eurojust στο δίκτυο συνεργασίας. δίκτυο συνεργασίας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει, θα συμπεριλαμβάνει και θα βασίζεται στις εργασίες που κάνουν μέχρι τώρα τα, ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των κρατών μελών για τους υπηρεσίες ασφάλειας του δικτύου. Κομισιόν και ενίσα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην οδηγία. Αν οι αρχές NIS εντός του δικτύου συνεργασίας ε, διαπιστώσουν ένα περιστατικό που φαίνεται να είναι εγκληματική ε, φύσης, θα πρέπει να ενημερώνονται η Europol. Οπότε η οδηγία συμπεριλαμβάνει έναν μηχανισμό στο να εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου και της NIS. ώστε να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το περιστατικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα κάνουμε και λεπτομερή συζήτηση. Θα είναι χρήσιμο να την παρακολουθήσετε κι εσείς. Δεν ξέρω, μήπω άλλοι συνάδελφοι θέλουν ε, να πούν τίποτε άλλο. Κυρία του, μήπως θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Απαντήσατε σημείο προς σημείο πολύ προσεκτικά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν ξέρω όμως για ένα θέμα, αν καταλάβατε καλά την ερώτηση που έχει θέσει ο Ανδρέας Σφάμπ. Για το διάλογο με τις τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει με ειδική εστίαση σε like-minded partners, σε εταίρους που έχουν τις ίδιες αξίες με μας. Αυτοί που έχουν όμως διαφορετική προσέγγιση που δεν έχουν τις ίδιες αξίες με μας, ε, τι θα κάνουμε με αυτούς. Το λέω γιατί νομίζω ότι δεν καταλάβατε πολύ καλά. Ναι, πράγματι δεν είχα καταλάβει πλήρως την ε, ερώτηση, αλλά κύριε Πρόεδρε, προτείνω να δώσω το λόγο στη συνάδελφο από την ΕΙΕΔ, να απαντήσει, αν θέλετε. Καλή ιδέα, πράγματι, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτη φορά μας θύμισε με την παρουσία του κάποιος από την ΑΕΔ για να μας ε, ε, πει οτιδήποτε, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εμένα που μου δίνετε το λόγο. Θα σας ε, εξηγήσω τη λογική πίσω από αυτό το διεθνές ε, σημείο που αφορά τη στρατηγή. Ο κυβερνοχώρος είναι ένας νέος τομέας ακόμα και για τους διπλωμάτες και για όσους ε, ασχολούνται με την προστασία των πιο σημαντικών πτυχών, ε, των πιο, σημαντικ, πιο σημαντικών ε, πιο σημαντικών στοιχείων κάθε κράτους μέλους και Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για το διάλογο με αυτές τις χώρες που δεν έχουν τις ίδιες αξίες με μας. Ο λόγος που το τονίζουμε όμως αυτό το θέμα στη στρατηγική είναι ότι θα θέλαμε αυτές ε, οι χώρες που δεν έχουν ακόμη καθορίσει ε, ποια είναι η θέση τους ακριβώς ε, στον κυβερνοχώρο. Θέλουν περισσότερη λογοκρισία στο ίντερνετ που είναι ένας ανοιχτός και ελεύθερος χώρος για την ώρα ή αν θα θέλανε να ευθυγραμμιστούν με μας για να διατηρηθεί το ίντερνετ ε, διαλειτουργικό και ελεύθερο. Ξέρετε ότι υπάρχει τεράστιος αγώνας στους διπλωματικούς κύκλους ε, για το θέμα αυτό, ε, τεράστια διαμάχη. Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αρχίσουμε με τους εταίρους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση. Πάντοτε πρέπει να έχουμε διάλογο και με ε, ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση, με, με χώρες που έχουν διαφορετική προσέγγιση, όπως την Κίνα για παράδειγμα, αλλά γι' αυτό ειδικά τον τομέα, τη στρατηγική ε, στον κυβερνοχώρο, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Και λέμε να αρχίσουμε με την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ε, Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις χώρες του ΩΣΑ, με την Αμερική, την Αυστραλία, με τις χώρες του Περιφερειακού Φόρου Μαζεάν, και επίσης προσπαθούμε να ε, οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και εκεί. Ο ΑΣΕ, συγγνώμη. Ε, όπως επίσης ε, προσπαθούμε να το ποινικό δίκαιο ε, να επικρατήσει γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που λένε ότι το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο που καλύπτει ε, και τις ε, περιόδους πολέμου πρέπει να, και αυτό πρέπει να αποτελέσει την έμπνευσή μας, ώστε να έχουμε αντίστοιχες, αντίστοιχους κανόνες και στον κυβερνοχώρο. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Απαντήσατε και στο ερώτημά μου. Εμένα με ενδιαφέρει και το θέμα της, ε, της προστασίας δεδομένων και την προστασία του ιδιωτικού βίου επίσης. Θα το γνωρίζετε, γιατί είμαι και εισηγητής για τέτοιο θέμα. Ένα πράγμα το οποίο ε, ενδιαφέρει πολύ το Κοινοβούλιο είναι ότι τα ζητήματα παραβίασης ασφάλειας, κατά πόσο θα έπρεπε να κοινοποιούνται ή όχι και αν θα έπρεπε να έχουμε κατεξιοδότηση πράξη. Όταν μας ήρθε η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε ρυθμιστική διαδικασία με παρακολούθηση ε, ήταν πολύ περίπλοκα τα πράγματα ήδη, όμως ε, είναι ακόμη πιο περίπλοκα τώρα γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω των ε, κατεξιοδότη συμπράξεων με το Συμβούλιο. Και επειδή έχω επιβιώσει πέντε τριμερών διαλόγων για το θέμα αυτό, για τα θέματα αυτά, των κατεξιοδότη συμπράξεων, γι' αυτό το λέω. Εγώ προτείνω να συμπεριλάβουμε τους κανόνες στη βασική πράξη και όχι να κάνουμε κατεξιοδότηση πράξης, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει μαζί μας. Ήταν μάλλον σχόλιο και λιγότερο ερώτηση. Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλαμε να έχουμε μια τέτοιου είδους ε, πράξη. Ε, δεν το είπαμε βέβαια τόσο σαφώς, αλλά πάση περιπτώσει είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε τη φύση της ε, πράξης. Ένα πολύ τελευταίο σημείο για αυτό το θέμα πάλι. Δεν θα σας εκπλήξει ότι οι χειριστές του δικτύου, οι φορείς παροχής ε, των ε, υπηρεσιών ε, αυτών είναι υπέρ του άρθρου 14 σε μεγάλο βαθμό. γιατί φυσικά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια του δικτύου τους και επίσης πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι, ισό, δεν είναι ίσος. Οπότε πραγματικά διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι εκείνοι διέπονται από τις ε, απαιτήσεις του άρθρου 13α, αλλά κάποιοι ε, άλλοι που ε, διεισδύουν στην αγορά με διαφορετικό τρόπο, μέσω των τηλεπικοινωνιών για παράδειγμα, δεν διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Um, Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και που απαντήσατε σε ερωτήσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, χρήσιμη ε, συζήτηση για να βασίσουμε τη δουλειά μας. Να ευχαριστήσω τον ε, Ανδρέα Σφάμπ, παρόλο που δεν είναι εδώ. Και τον κύριο Γκαρσέ Ραμόν επίσης για τα σχόλιά του. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης, αλλά και τις εργασίες μας για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίασή μας ε, θα είναι 7 Μαΐου, 9 με 12.30. Έκτακτη συνεδρίαση και μετά η επόμενή μας ε, συνεδρίαση νομίζω 27 Μαΐου. Θα έχουμε δύο γεμάτες μέρες και το Μάιο. Ελπίζουμε να μας ξαναπαρακολουθήσετε κι εσείς στο διαδίκτυο. 29 με 30 Μαΐου διορθώνει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Είναι ηλιόλουστο το απόγευμα. Βλέπω ότι σιγά σιγά φεύγετε. Πηγαίνετε προς την πλατεία Λουξεμβούργου. Οι περισσότεροι θα φύγετε, αλλά εμείς ε, που δουλεύουμε για τις ε, παραγορήσεις και τον τριμερή διάλογο θα πρέπει να παραμείνουμε. Ευχαριστώ πολύ πάντως.